Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω τις εργασίες εν αναμονή των υπόλοιπων συναδέλφων. Ε, αν υπάρχουν ε, διαφωνίες θα δούμε τι θα κάνουμε. Στο πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη έχουμε την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης που σας έχει διανεμηθεί. Υπάρχουν ενστάσεις για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 15ης και 16ης Μαρτίου του 2011. Ενστάσεις. Ωραία. Περνάμε στο σημείο υπαριθμών 3. για τις εργασίες αυτών των δύο συνεδριάσεων. Να σας πω ότι κατόπιν επαφών με τους αναφέροντες, το σημείο 24 θα γίνει ε, μετά το σημείο 12, τα σημεία 10 και 11 αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση. Είναι παρόντες οι αναφέροντες για τις αναφορές που έχουμε στα σημεία 16, 12, 16 και 21 και πιο συγκεκριμένα για την αναφορά 575 του 2010 να σας επισημάνω ότι θα υπάρξει και μία παρέμβαση με την προβολή ενός σύντομου φιλμ διάρκειας περίπου δύο λεπτών. Όσον αφορά τώρα το σημείο υπαριθμών 15, οι αναφέροντες θα παρακολουθήσουν τη συζήτησή μας μέσω web streaming από τη Μάλτα. Και για την αναφορά που έχουμε στο σημείο 25, ο κύριος Μίτσελ ζήτησε να διαβάσει στην αίθουσα μία δήλωσή του για, την, ε, ε, για τον απορροφερετήρα του Πούλμπερκ στον κόλπο του Δουβλίνου. Όπως και σε κάθε συνεδρίωση έχετε λάβει και το παράρτημα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνει και τις ενδείξεις για τις αναφορές τις οποίες θα περατωθούν με γραπτή απάντηση. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το πέρας των ε, συζητήσεων στη συνεδρίασή μας ε, θα ακολουθήσουμε την πρόταση που έχει διατυπωθεί από τη γραμματεία. Να περάσουμε τώρα λοιπόν στο σημείο 5. Περνάμε στα ουσιώδη πλέον. Αναφορά παριθμό 1594 του 2010 από τον κύριο Γκαμπριέλε Τσέρβι. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, επομένως δίνω απευθεία το λόγο στον κύριο William Floyd από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε από τα πρόσφατα αποτελέσματα από το δικαστήριο στο Στρασβούργο, η αναφορά αυτή φαίνεται ότι έχει πλέον ε, ικανοποιηθεί. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν αντίστοιχο θέμα, διότι υπήρξε και προφορική ερώτηση με συζήτηση για το θέμα αυτό το Νοέμβριο του 2009 στην Ολομέλεια και όπως ε, θα θυμάστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυστυχώς είχε επισημάνει ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα της Ιταλίας και δεν υποχρεώται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση επί του θέματος. Θεωρήσαμε ότι πρόκειται για εθνικό ζήτημα και συνεπώς ε, ο αναφέρον ακολούθησε την ε, σωστή διαδικασία και έκανε έκκληση στο εφετείο και πήγε στο δικαστήριο στο Στρασβούργο, το οποίο εξέδωσε τώρα και απόφαση. Κύριε Όκεν. Με εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά εδώ. Δεν ήξερα ότι μπορεί κάποιος να υποβάλει αναφορά για απόφαση δικαστηρίου. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές με τις οποίες ε, διαφωνώ συνήθως ε, και διαφωνώ και με το αίτημα και εδώ με εξέπληξε το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια υπόθεση η οποία ήταν υπόθεση δικαστηρίου. Καταλαβαίνω τη δική σα θέση, δεν τα έχω μαζί σα, αλλά γιατί συζητάμε εμείς στην ημερήσια διάταξή μας μια τέτοια αναφορά. Με εκπλήσει πραγματικά μία υπόθεση που έχει αποτελέσει δική μου συζήτηση στο δικαστήριο, είτε αποφάσισε είτε όχι και τώρα ξανασυζητάτε στο δικαστήριο, δεν θα επισέλθω στην ουσία, δεν είναι αναφορά. Είναι αναφορά γιατί κάποιο ε, τη δηλώνει ω αναφορά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πάρα πολλέ που θεωρούνται μη παραδεκτέ, αλλά δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ σε εμά με απόφαση δικαστηρίου, στο Στρασβούργο κιόλα. Ή μπορούμε, μπορεί κάποιος ε, από εμά ε, να ε, αμφισβητεί την απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση. Ο κύριος Γιάρ. Ε, δεν με βλέπετε ίσως γιατί είναι μπροστά μου το καρσόνι αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό γιατί αυτή η διαφορά υπάρχει πάντοτε. Υπάρχουν αναφορές τις οποίες συζητάμε, μένουν αναχτές και όπου ενδεχομένως ο αναφέρον μπορεί να απευθυνθεί και στα δικαστήρια. Κάποια στιγμή λοιπόν το δικαστήριο αποφασίζει είτε υπέρ είτε κατά της αγωγής και μετά μπορεί να επανέλθει εδώ η αναφορά. Οπότε ε, ενδέχεται να είναι αυτός ο λόγος ε, βάσει του οποίου έχει αποφασίσει σωστά και ε, η Επιτροπή μπορεί ίσως να ξανασυζητήσει αν η νομοθεσία είναι σωστή είναι κάτι το οποίο ίσως μπορούμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και να πούμε ότι θα κλείσουμε αυτό το θέμα αυτής της αναφοράς και μετά να συζητήσουμε από της ουσίας. Στο 5 ε, πρέπει να σας πω ότι αποφάσισε ε, το, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά εγώ δεν βλέπω γιατί εδώ πρέπει να αποκλείσουμε τη συζήτηση αυτής της αναφοράς είμαστε ένα πολιτικό όργανο, δεν είμαστε δικαστήριο, άρα μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς ε, βάσει πολιτικών κριτηρίων πώς θέλουμε να κινηθούμε. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι μπορούμε και σε αυτό το σημείο να κλείσουμε την, ε, την αναφορά αυτή. Συναδελφοί, παρακαλώ, κύριος Βίλαντ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στην κυρία Όκεν ότι αποκλειστικά και μόνο με το γεγονός ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, που είναι ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί να δικαιώσει ή όχι τον αναφέροντα δεν είναι λόγος για να μην δεχθούμε μία ε, αναφορά να μην τη θεωρήσουμε παραδεκτή. Το θέμα είναι ότι ε, είτε θα βασιστούμε στην νομοθεσία είτε στην ε, ε, απόφαση του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Αλλά ε, μπορεί ίσως το, μπορεί το θέμα να συνάδει με την νομοθεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά εμείς παραδείγματος χάρη μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι παραδεκτή μία αναφορά. Δηλαδή ακόμη και αν έχει βγει, εκδοθεί δικαστική απόφαση για μία αναφορά μπορεί να επανέλθει εδώ το θέμα και να αποφασίσουμε αν εμείς θέλουμε να κλείσουμε την αναφορά ή να την κρατήσουμε ανοιχτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είπαμε ότι πρέπει να κλείσει. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση όμως σε όλους τους συναδέλφους, διότι Καταρχήν, συμφωνώ με τις απόψεις που εξέφρασε η συνάδελφος Άουκεν. Ως προς την ουσία όμως ε, δεν έχουν ε, ε, σχέση με το αυτό που συζητάμε, αλλά εμείς συζητάμε την επαύριο μίας απόφασης που μόλις εκδόθηκε. Η αναφορά όμως παρουσιάστηκε από τον αναφέροντα διότι θεωρούσε ότι δεν συνάδει με τις θεμελιώδεις αρχές από τις οποίες εμπνέονται οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα έπρεπε να υπάρχει ε, υποχρέωση να ε, κατέβουν σταυρωμένοι από τα Ιταλικά σχολεία. Εμείς γι' αυτό τη δεχτήκαμε. Υπήρξε και κρεμότητα για το δικαστήριο. Ως συνήθω ε, αναβάλαμε την αναφορά και σήμερα την ξαναβάλαμε στην ημερήσια διάταξη για να πούμε ότι η αναφορά συγκεκριμένη έχει κλείσει διότι εμείς είχαμε αναβάλει την απόφασή μας για να ακούσουμε την απόφαση του δικαστηρίου και το δικαστήριο εξέδωσε μία απόφαση που Έχετε αυτή την υπόθεση παραβίαση δικαιωμάτων. Αυτή τη στιγμή υποχρεώνει την Ιταλία να μην διατηρήσει πλέον του εσταυρωμένου στα σχολεία. Ε, αυτό για να μην ε, κάνουμε συζήτηση από λανθασμένο σημείο. Μισό λεπτό και θα συνεχίσουμε. Κυρία Όκεν, ε, έχουμε και άλλους συναδέλφου που θέλουν να μιλήσουν. Η κυρία Μπιτζότο θέλει το λόγο και μετά θα σας ξαναδώσω το λόγο. Η κυρία Μπιτζότο δεν θα μιλήσει. Η κυρία Όκεν. Απλά να πω ότι συμφωνώ ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Είναι λίγο περίεργο γιατί εμείς δεν φτιάχνουμε τους νόμους σε αυτή την Επιτροπή εδώ. Και αν έχεις το ανώτατο δικαστήριο, ακόμα και αν διαφωνείς και εγώ πιστεύω, είμαι χριστιανή και είμαι υπέρ της πρώτης απόφασης, διότι ε, νιώσα πολύ άβολα όταν ε, αποκαλέσαμε σύμβολο των εσταυρωμένων. Είναι κάτι παραπάνω από σύμβολο, πολύ περισσότερο. Ε, έχω διαφορετική θέση και είμαι σύμφωνη με την πρώτη απόφαση, διότι αυτό είναι πολύ ισχυρό σύμβολο και μήνυμα ο εσταυρωμένος. Αλλά τώρα θέλω να θυμηθούμε ότι δεν είναι μόνο όταν είναι πολιτικό, σβολικό για κάποια ε, κόμματα που βρίσκονται εδώ και τότε αποδεχόμαστε ε, αναφορές ε, για ανθρώπινα δικαιώματα. Εάν, ε, δεν πρέπει να πούμε ότι αυτό αφορά χριστιανικές ιταλικές αξίες, θα το πάρουμε, αυτό αφορά κάτι άλλο, δεν θα το δεχτούμε. Αυτός είναι ο κίνδυνος κατά την άποψη ε, ε, όλοι έχουν πει ότι ωραία θα το δεχτούμε ως αναφορά. Ωραία. Τώρα αυτός είναι ο κανόνας και η διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά να προσθέσουμε ούτως ή άλλως. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συγκεκριμένη αναφορά Έκλεισε και περνάμε στο επόμενο σημείο. Αναφορά υπαριθμών 901 του 2008 που παρουσιάζει ο κύριος David Skinner, ο οποίος είναι παρόν και του δίνουμε το λόγο για τρία λεπτά. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε, έχει ήδη γίνει δύο φορές συζήτηση για αυτή την αναφορά εδώ και έχει μεγάλο ενδιαφέρον από βουλευτές και σε αυτή την Επιτροπή και εκτός αυτής. Ε, έχει, ε, έχει μεγάλη υποστήριξη. αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω ποιο ακριβώς είναι το θέμα. Και θα ήθελα να φυστήσω ε, την προσοχή σε δύο τύπους ελευθερίας του συνεταιρίζεσθε. Υπάρχει το θετικό και το αρνητικό δικαίωμα. Το αρνητικό δικαίωμα ορίζεται ως η ελευθερία από την παρέμβαση από άλλους ανθρώπους που θέλουν να ε, συνεταιρίζεστε μαζί τους και έρχεται σε αντίθεση με το θετικό δικαίωμα που ορίζεται ως η ελευθερία ενός ατόμου να συνεταιρίζεστε με αυτούς που αυτός επιθυμεί. Αυτή η διάκριση είναι βαθιά ενσωματωμένη στην κοινωνία μας, στους πολιτισμούς μας, σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε και νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν ότι ένα αρνητικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο δικαίωμα. Ένα αρνητικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε είναι ένα απόλυτο δικαίωμα και χρήζει προστασίας. Αυτή η αναφορά που υποβάλαμε το 2008 ήταν αποτέλεσμα μια σειράς από εργασιακές συγκρούσεις στην Σουηδία το 2006. Και τώρα έχουμε ε, τεκμηριώσει ότι τα άτομα πρέπει να έχουν την ελευθερία να επιλέγουν να μην υπογράφουν μια συλλογική σύμβαση και να επιλέγουν να μην συμμετέχουν σε ένα συνδικάτο όπως το έχω πράξει. Ένα μέλος αυτής της Επιτροπής μας είπε πρόσφατα και παραθέτω εάν θέλω να απολαμβάνω την ελευθερία του συνεταιρίζεσαι τότε πρέπει να είμαι σε θέση να απολαμβάνω και την ελευθερία του να μην συνεταιρίζομαι. Άρα ε, πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Και αυτή, αυτός είναι ο πυρήνας της αναφοράς μας και γι' αυτό είναι το σημαντικό να δώσει συνέχεια η Επιτροπή σε αυτή. Δεν συζητάμε το γιατί κάποιος δεν διαπραγματεύεται με τα συνδικάτα ή ποιοι είναι οι λόγοι του. Το θέμα είναι ότι αυτό το άτομο έχει απόλυτο δικαίωμα να πει όχι στις διαπραγματεύσεις. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ε, μέλη εδώ που θα λέγανε και τι έχετε να πείτε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα, εργαζομένων, τα δικαιώματα των ε, συνδικάτων. Αυτά δεν παραβλέπονται, δεν δεν προβλέπονται. Υπάρχουν και εκεί βασικέ θεμελιώδει ελευθερίες, αλλά θέλουμε να θεωρήσετε το εξή. Εάν ένας εργοδότη δεν έχει εργαζόμενους σε συνδικάτο και αυτός ο εργοδότη πληρώνει μισθού, που είναι καλοί ή καλύτεροι από αυτούς που ζητά το συνδικάτο και δεν υπάρχει λογική βάση για τα συνδικάτα να προσπαθήσουν να ξαναγκάσουν την εταιρεία να υποβληθεί σε αυτή αλλά να παίρνει δράση που πιστεύω ότι είναι απαραίτητη αυτό είναι άρνηση της αρχής της ελευθερίας της, του μη συνεταιρίζηση και διάκριση κατά του δικαιώματος. Πιστεύουμε ότι δεν είναι αποδεκτό στην Σουηδία και σε άλλα κρατημέλη το εθνικό ε, δίκαιο, το εργατικό δίκαιο να μην προβλέπει για ε, την ύπαρξη ενός συστήματος διαπραγμάτευσης που να είναι δίκαιο και ισορροπημένο ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Πολλοί εργοδότες δεν θέλουν να, πολλοί εργοδότες δεν θέλουν να είναι μέλη ε, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε συνδέσμου, θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, να έχουν τη δική τους επιχείρηση και Υπάρχουν και εργοδότες και εργαζόμενοι που έχουν πολύ έντονες πεπιθήσεις για το θέμα αυτό και έχουν μικρές επιχειρήσεις που στηρίζονται σε εξαιρετικές και δίκες σχέσεις στο χώρο εργασίας. Αλλά αυτό που ζητούν και αυτό που αναμένουν είναι όπως οι κυβερνήσεις να είναι διατηθειμένες να τους παρέχουν μια αξιοπρεπή προστασία από τον εξευτελισμό ε, των ε, συνδικάτων που θέλουν να δείξουν ότι είναι τα ισχυρότερα στην αγορά εργασίας. Σήμερα η οικονομική οικονομική κρίση και η υψηλή ενεργεία θα πρέπει να μας δείξουν ότι η Ευρώπη χρειάζεται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, χρειάζεται τους επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και εταιρείε με ευελιξία, και χρειάζονται ε, την ευκαιρία να σταθούν στα πόδια τους και να μην υποβάλλονται σε απειλές χωρίς δικαιολογία από κάποιον οργανισμό που ε, δεν έχει κανένα ενδιασμό στο να τους κλείσει αν αρνηθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους. Για ε, τόσο καιρό πιστεύαμε ότι αυτή η ελευθερία είχε μόνο θετική εφαρμογή αλλά είναι σαφές ότι τα άτομα έχουν και ένα καθοριστικό δικαιώμα να επιλέγουν να μην συμμετέχουν. Και δεν μιλάμε μόνο για το και για την αρχή των συλλογικών συμβάσεων μιλάμε για μια αρχή της ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσαι, μια βασική θεμελιώδη ελευθερία. Ε, ευχαριστούμε τους ε, πολλούς βουλευτές που έχουν ε, υποστηρίξει και έχουν επιδείξει το ενδιαφέρον τους και ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει επιθυμία εκ μέρους αυτής της Επιτροπής να παραπέμψει στο Κοινοβούλιο ε, και θα θέλαμε, κυρία Πρόεδρε, αν ε, θα μπορούσατε να διορίσετε έναν εισηγητή, διότι αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα στα μέλη εν ώψη της ε, σύνταξης μιας μη νομοθετικής έκθεσης. Θα θέλαμε να προχωρήσετε, κυρία Πρόεδρε και μέλη, με, αυτή την, με αυτές τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο ε, για άλλη μια φορά να υποστηρίξει τα βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και να υπερασπίση της ελευθερίας όλων των πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον κύριο Σένστρ. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος διότι ήδη πολλά ελέγχθησαν στις δύο προηγούμενες ευκαιρίες και θα ήθελα απλώς να πω εις τους ευρωβουλευτές και μέλη αυτής της Επιτροπής ότι όσο ατυχές και να είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση Γκούσταυσον που ήταν μια περίπτωση για αναθεώρηση αποφάσισε ότι το επίπεδο της συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε δεν ε, είναι νόμος και ε, αυτό είναι το, ε, συνάδει με την απάντηση της Σουηδικής κυβέρνησης σχετικά με την Σουηδική περίπτωση και δεν χρειάζεται να σχολιάσω περαιτέρω σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Σέλνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ αισθάνομαι ότι αυτά τα έχω ξανακούσει και ξαναδεί διότι έρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και πριν από πολλά χρόνια, πριν από 25-30 χρόνια έγινε μια μεγάλη συζήτηση για αυτό που λέμε αγγλικά τα ε, closed shops, δηλαδή όπου ε, ήταν υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να συμμετάσχει σε μια συνδικαλιστική οργάνωση και τότε επί κυβερνήσεως Θάτσε απεφασίστη να καταργηθούν τα closed shops και να υπάρχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ή μη. Δηλαδή να γίνει κανείς ή να μην γίνει μέρος μιας συνδικαλιστικής οργανώσεως χωρίς αυτό να συνεπιφέρει υποχρεώσεις που μπορούν να τους επιβληθούν από την επιχείρηση όπου εργάζονται και ε, γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ απλούστατα επανερχόμαστε στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου που υπήρχε τότε και το δικαίωμα συνεταιρίζεστε ή μη ε, έχει Εδρεωθεί σε διάφορους χάρτες επί δεκαετίες. Ε, μπροστά μου έχω την ε, Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίων Δικαιωμάτων και στο άρθρο 20 λέγεται ότι ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα ελεύθερη συγκεντρώσεως και συνεταιρι... του συνεταιρίζεστε χωρίς όμως να είναι κανείς υποχρεωμένος να συνεταιριστεί. Υπάρχουν τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων που υιοθετήθηκαν το Δεκέμβριο του 1989 και ίσως η Επιτροπή αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο, αναφέρθηκε όμως στο άρθρο ή στην παράγραφο 11 και εγώ τώρα θα επαναρχόμουν στο, συμπαράγραφο παράγραφο ή άρθρο 11 που λέγεται ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έχουν δικαίωμα να συνεταιρίζονται εντός συνδικαλιστικών οργανώσεων ή ε, ενώσεων και επιπλέον ότι ο κάθε εργοδότης μπορεί να συμμετάσχει ή μη σε μια τέτοια οργάνωση χωρίς ε, να χρειαστεί να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να είναι πιο συγκεκριμένος διότι το δικαίωμα των, των εργαζομένων να συνεταιριστούν ή όχι εδρεώνεται και από την διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την διακήρυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και 20 χρόνια μετά ερχόμαστε εδώ σε μια συζήτηση να διαφωνούμε εάν μπορούν να εφαρμοστούν εφαρμοστούν αυτά τα δικαιώματα των εργαζομένων, πράγμα το οποίο βρίσκω περίεργο. Θα έλεγα λοιπόν ο αναφέρον και η Επιτροπή να συμφωνήσουν να υπάρξει μία προφορική ερώτηση επί του θέματος και εγώ θα στήριζα την πρόταση ε, του αναφέροντα να υπάρχει ένας συζητητής επί του θέματος που είναι βασικό θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ε, εδρεώνεται μέσω της ε, παγκόσμιας διακηρύξεως και του χάρτη και ισχύει πέραν των 20 ετών. Η κυρία Όκεν. Να πω απλώς ότι Διαφωνώ απολύτως με το συνάδελφο. Και το λέω διότι και πάλι αφού έχουμε απόφαση από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όπω κάναμε και στην Ιταλική περίπτωση, μπορεί να προσπαθήσουμε να ξαναπροσφύγουμε στο δικαστήριο, αλλά δεν είναι δική μα αρμοδιότητα και μάλιστα σε ένα τομέα για τον οποίο δεν υπάρχει νομοθεσία στην Ευρώπη. Δεν είναι δική μα ε, η νομοθεσία. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε εδώ στην Επιτροπή. Θεωρώ ότι είναι κατασπατάληση του χρόνου μας να καθόμαστε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που καθόμαστε εδώ και το συζητάμε. Ε, μπορεί να συμφωνούμε, να διαφωνούμε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα, αλλά υπάρχει απόφαση και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα όσα συνέβησαν. Μπορεί κάποιο να ξαναπροσφύγει στο δικαστήριο, όπω έγινε και με την περίπτωση της Ιταλίας, αλλά δεν είναι δική μα δουλειά. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά εδώ στην Επιτροπή μας. Μπορεί να μας ενδιαφέρει να μην έχουμε το σουηδικό, δανέζικο μοντέλο και να λέμε ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, παρόλο που λέτε ότι δεν είναι αυτό, αυτό είναι. Εγώ δεν μπορώ να προασπίσω το δανέζικο ή το σουηδικό μοντέλο ε, καθυστερώντας εδώ την Επιτροπή ή να το υποσκάψω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να συζητάμε τώρα εδώ με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν είναι δική μας δουλειά. Αυτή είναι η θέση μου. Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Σπανίως συμφωνώ με τον Ρότζερ Χέλμερ, αλλά δυστυχώς το ένστικτό μου σε αυτή την περίπτωση μου λέει ότι μάλλον έχει δίκιο χρησιμοποιείται καταπιεστικός μηχανισμός ε, στη Σουηδία και χρειάζεται περαιτέρω εξέταση ε, αν μπορούμε να το πετύχουμε. Ο κύριος Γιάρο. Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ του να γίνει μία προφορική ερώτηση αλλά πιστεύω ότι το κάθε κράτος μέλος έχει κάποιο σκεπτικό. Δηλαδή δεν θέλουμε εδώ να αποφασίσουμε επιθεμελιωδών δικαιωμάτων. Εάν κάποιος θέλει να συνεταιριστεί, εάν θέλει να καταρτήσει μία οργάνωση και να γίνει μέλος, ε, είναι δικαίωμα αλλά δεν είναι κατανανταστικό. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε με διάφορα ε, παρεμφερή παράπονα στη Γερμανία μπορεί κανείς, δεν μπορεί κανείς να αποτελέσει μέλος μιας οργάνωσης χωρίς να έχει ερωτηθεί. Ε, υπάρχουν δηλαδή νομικές διαφωνίες επί αυτού και όσον αφορά το, την αρνητική αρχή της ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσαι είναι κάτι που θα έπρεπε να συζητήσουμε διότι εδώ είναι ότι επιβάλλουμε σε ορισμένες ομάδες δικαιώματα που δεν ζήτησαν για κάθε έναν, για κάθε συμπεριφορά η οποία φαίνεται παράλογη μπορεί να υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη αλλά ε, εάν η κοινωνία δεχθεί μία αρνητική ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε, τότε θα συμφωνούσα να υποβληθεί μία προφορική ερώτηση, να εξεταστεί και να έχουμε μία έγκυρη απάντηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται εδώ να εμπλέξουμε τα κράτη-μέλη, αλλά βρίσκω μάλλον περίεργο ένα άτομο το οποίο δεν έχει ερωτηθεί υποχρεωτικά να ανήκει σε μία οργάνωση. Δηλαδή ποια είναι η αιτιολογία αυτό δεν συνάδει με την δημοκρατία και το κράτος δικαίου είναι υποχρεωτικός σοσιαλισμός διότι ε, σήμερα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχουμε πολλά παράπονα τέτοιου είδους ιδίως από εργαζομένους οι οποίοι θεωρούν ότι συμμετέχουν σε επιμελητήρια, σε οργανώσεις, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς να έχουν ερωτηθεί και θεωρούνται ότι όντως είναι μέλη τους. Υπάρχει λοιπόν πρόταση για προφορική ερώτηση. Ο κύριος Σκίνερ για δύο λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ το γεγονό ότι μου δίνετε το λόγο. Ο κύριο Φίνστρεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανέφερε την απάντηση τη ειδική κυβέρνηση προ εσά. Αν διαβάσετε όμω τι γράφει ο κύριο Λιτερίν, ο Υπουργό Εργασία τότε, λέει στην απάντησή του ότι δέχεται την αρχή της, αρνητικής, της ελευθερίας του συνεταιρίζεστε. Η Σουηδική κυβέρνηση δέχεται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η Επιτροπή σας είναι η αρμόδια για να συζητήσει κατά πόσον η Σουηδική εργατική νομοθεσία παραβιάζει αυτή την ελευθερία. Ο Υπουργό τη δέχεται και επομένω δεν μπορεί ο κύριο από την Επιτροπή να μα λέει ότι δεν υπάρχει αρνητική ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Ακόμα και η Σουηδική κυβέρνηση δέχεται ότι υπάρχει και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητάται ακόμα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο και αυτό το γνωρίζω, είναι γεγονό. Ευχαριστώ. Πράγματι, στο σημείωμα που λάβαμε από την Σουηδική κυβέρνηση υπάρχει αυτή η διευκρίνηση και εδώ θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο δεν είναι δευτερευούση σημασία. Η απόφαση αυτή η οποία αναφέρθηκε επανειλημμένως από το δικαστήριο και αναφέρεται και στα έγγραφά μας Καταρχάς δεν είναι μία απόφαση που αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση που συζητάμε και κατά δεύτερον ο λόγος ο οποίος παρουσιάζεται ως σύννεψη στα έγγραφά μας σε καμία περίπτωση δεν απαντά σε αυτό το οποίο απασχολεί εμάς. Διότι πρόκειται για μία απόφαση που αφορά απλώς και μόνο το πώς έχει την νομοθεσία. Και το δικαστήριο λέει πράγματι στη Σουηδία δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα του μη συνεταιρίζεστε. Πρόκειται για μία δήλωση η οποία δεν έχει καμία σημασία εάν δεν εξετάσουμε περαιτέρω το περιεχόμενο της απόφασης. Και ούτως ή άλλως ε, την απορρίπτει ο ίδιο ο υπουργό, ο οποίος δηλώνει ότι το δικαίωμα του μη συνεστερίζεστε είναι ένα δικαίωμα το οποίο μπορεί να ασκήσει κάποιο ελεύθερο. Να παρουσιάσω εδώ και τη δική μου την άποψη. Νομίζω ότι σας την έχω πει και στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη αναφορά ακολούθησε μία περίεργη οδό. Ε, δεν έλαβε τη δέουσα προσοχή και δεν δόθηκαν οι δέουσες απαντήσεις, διότι το να διεκδικεί κάποιος ε, το δικαίωμα του μη συνεταιρίζεστε και την ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε, το έχουμε συσχετίσει και με την, ε, ε, το γεγονός ότι έχει σχέση με θρησκευτικού λόγους. Αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο που θέλησε να δώσει ο αναφέρον μαζί με κάποιους άλλους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά το γεγονός είναι ότι μας ζητάτε να αξιολογήσουμε εάν παραβιάζονται οι αρχές οι οποίες έχουν εγγραφεί στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελευθερία του μη συνεταιρίζεστε ε, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον είναι αρχή και κατά πόσον αυτή η αρχή παραβιάζεται από τους ειδικέ αρχέ ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε το θέμα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσον είναι αναρμόδια η Επιτροπή μας όταν έχουμε συζητήσει επανελειμμένως το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά τώρα το αίτημα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει μέσω προφορικής ερώτησης. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα αιτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι αντίθετος σε αυτό το αίτημα ή μπορούμε να κλείσουμε το σημείο με την απόφαση αυτή. Θα μπορούσα να ρωτήσω τους αδέλφους. Συμφωνούμε όλοι. Η κυρία Όκεν διαφωνεί. Θέλει το λόγο. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια της κυρίας Όκεν. Δηλώνει ότι είναι κατά μάλλον η κυρία Όκεν, αλλά συγγνώμη δεν ακούμε. Νόμιζα ότι θέλετε το λόγο, κυρία Όκεν. Η κυρία Όκεν, ρωτήσατε αν είναι κάποιος κατά και είπα ναι, εγώ είμαι κατά. Συγγνώμη κυρία συνάδελφα. Νόμιζα ότι ζητούσατε το λόγο και σας είπα μισό λεπτό. Ολοκληρώνω. Λοιπόν, έχετε αντίρρηση λοιπόν. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχουμε πλειοψηφία για το συγκεκριμένο αίτημα και κλείνουμε την αναφορά προς το παρόν, μάλλον το σημείο αυτό προς το παρόν και αποφασίζουμε να παρουσιάσουμε προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Είμαστε στο σημείο 7 ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών και θα ήθελα να δώσω απευθείας το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μέγερ, για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψε στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη γραμματεία μου λένε ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορούμε να έχουμε το πρώτο σχέδιο έκθεσης, το οποίο θα προκύψει από τις ε, πρώτε ανταλλαγέ απόψεων που κάναμε στο θέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα να σας ζητήσω είναι το εξή. Την επόμενη εβδομάδα όταν θα έχουμε το σχέδιο έκθεσης, και οι σκιώδει εισηγητές ε, θα έχουν το σχέδιο, θα ήθελα να το μελετήσουν και να κάνουμε μία συνεδρίαση με τους σκιώδει ε, στις αρχές Μαΐου έχοντας όλοι διαβάσει τα μαθήματά μας ε, και να έχει ο καθένας και τις ε, προτάσεις του από πλευράς πολιτικών ομάδων ε, για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση για το πρώτο έγγραφο και να έχουν όλες οι ομάδες εκφράσει την άποψή τους. Αυτό προτείνω. Συμφωνείτε? Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ. Ευχαριστώ να ρωτήσω τον κύριο Μάιερ, μήπως θα γίνει συζήτηση σήμερα, έχετε πρόθεση να κάνουμε, συζήτηση για αυτό το σχέδιο που έχουμε μπροστά μας. Ε, ρωτώ γιατί μου ζητήθηκε από την Άλτε να είμαι σκιώδης για το θέμα αυτό, που με τα χαρά θα το κάνω. Ε, λοιπόν, η πρότασή μου θα ήταν είτε να επενδυθεί σαν ερώτηση ή να ρωτήσουμε τον κύριο Μάγερ αν δεν μπορεί να οργανωθεί μία συνεδρίαση σκιωδών και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την συνεδρίαση για την επόμενη φορά μεταξύ σκιωδών εισηγητών κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε την Επιτροπή καλύτερα. Κύριος Μέγερ. Ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το μόνο που σας είπα είναι ότι η γραμματεία μπορεί να παρουσιάσει ένα πρώτο σχέδιο κειμένου και ότι όλοι οι σκιώδη συζητητές ε, θα λάβουν το έγγραφο αυτό την επόμενη εβδομάδα και κατόπιν, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των σκιωδών εισηγητών, θα γίνει μια συνεδρίαση του εισηγητή με όλους τους σκιώδεις και εκεί θα ετοιμάσουμε το έγγραφο το οποίο όλοι και όλες συμφωνούμε ότι είναι το έγγραφο το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουμε στην Επιτροπή. Πρόεδρος, νομίζω ότι συμφωνείτε όλοι. Θα συνεννοηθεί ε, ο εισηγητή με τους ε, σκιώδει και στην επόμενη συνεδρίαση θα παρουσιάσουμε και ένα σχέδιο έξοδο. Έκθεση, συγγνώμη. Επόμενο σημείο η συζήτηση ε, για την κινητικότητα και την ένταξη, αλλά απουσιάζει ο κύριος ε, Τσίτσεστερ. Μήπως έχω κάνει λάθος. Είναι εδώ ο κύριος Τσίτσεστερ. Να ζητήσω από τη συνάδελφο Άουκεν αν μπορούμε να συζητήσουμε το δικό της σημείο, τη γνωμοδότηση για την 27η ε, ετήσια έκθεση της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να δώσω το λόγο στην κυρία Άουκεν για το σημείο 9.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 Δεν θέλω να υπησέλθω σε όλα τα θέματα, αλλά ουσιαστικά να τονίσω μόνο τα βασικά σημεία, δηλαδή το σημείο 3 του σχεδίου. πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί από τους ετούντες έρχονται και ε, νομίζουν ότι ισχύει ο χάρτη και εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο σχετικά με τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Ίσως λοιπόν καλό θα ήταν να εξετάσουμε εις βάθος το θέμα και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και έχουμε δύο καλά παραδείγματα εδώ όπου πραγματικά εξετάζουμε τα δικαιώματα και αναφέρομαι στα δύο πρώτα θέματα τα οποία συζητήσαμε και ε, υπάρχει η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η οποία θα επιθυμούσε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Στην ε, απάντησή μας θα ζητήσουμε από τις εθνικές αρχές, δικαστικές αρχές να αποφανθούν. Διότι ε, σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένες πόλεις, στην Ισπανία, σε ε, θέματα παγκοσμιοποίησης ε, ίσως ε, οι αναφέροντες ζητήθηκε από τους αναφέροντες να στραφούν στα εθνικά δικαστήρια και μας είπαν μα αυτοί έχουν πάρα πολλή δουλειά, δεν θα τα επεξεργαστούν και το, ή το κόστος είναι τόσο υψηλό ώστε δεν μπορούμε εμείς να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς σωστά την ε, εφαρμογή της νομοθεσίας και είδαμε ότι εδώ μιλάμε για 2.900 ή 3.000 παραβιάσεις ακόμη και αν αριθμητικά μειώνονται είναι πάρα πολλές οπότε μπορεί να πούμε ότι ίσως αριθμητικά μειώνονται ε, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικές και κοιτάζω τα έγγραφά μου οπότε διαπιστώνω ότι η νομική επιτροπή ζητεί όλα αυτά να γίνουν νόμιμα ε, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν ε, είναι τυχαίο ότι ασχέτως του αν ένα θέμα ε, τίθεται για πρώτη, δεύτερη, δέκατη φορά θα πρέπει να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη διαδικασία και θα πρέπει σήμερα να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ε, στην διαδικασία αυτή την οποία μας ζητά η νομική επιτροπή. Όσον αφορά το 5 και το 10 είναι σημαντικά διότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πολύ αργά την ε, οδηγία και το ίμιση των αναφορών αναφέρεται σε αυτό το θέμα διότι καταρχήν ε, αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα εάν έχουμε περίπλοκους νόμους με πολλούς αριθμούς και στη συνέχεια τα κράτη αδιαφορούν και δεν αντιδρούν εγκαίρως. Δεν είναι ικανοποιητική δηλαδή αυτή η διαδικασία. Τώρα, σχετικά με το σημείο 3 της εκθέσεώς μου, μάλλον το 12, ε, που έχει σχέση ε, με το 3 δηλαδή του πότε τα θέματα εξετάζονται. Εγώ δεν ξέχνω ότι ε, έχουν αποδεσμευτεί διάφορα από αυτά τα θέματα και στη συνέχεια βλέπουμε ότι μπορεί κανείς να παραβιάσει τα θέματα αυτά ε, ή να στραφεί προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Γι' αυτό και η Επιτροπή στο σημείο αυτό πρέπει να τοποθετηθεί σχετικά με αυτό το πρόβλημα διότι ουσιαστικά πολλές από τις αναφορές ε, άπτονται αυτού του θέματος ε, και γι' αυτό και προσφάτως όταν συζητούσαμε το άρθρο 7 σε σχέση με το άρθρο 2 είπαν ότι αυτό ήταν μια ατομική βόμβα. Βεβαίως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσει κανείς ατομικές βόμβες. Δεν υπάρχει καμία διάταξη η οποία να έχει επιρροή ατομικής βόμβας, αλλά εδώ έχουμε διάφορες δυνατότητες αντίδρασης και μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά να αποφασίζουμε τι θα πράξουμε και αυτή η ευέλικτη απόφαση ε, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και τέλος, υπάρχει το θέμα της ε, διαφανείας. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δίκιο. Και ότι σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε ε, να ε, τοποθετηθούμε και να αποφανθούμε επί μίας γραπτής αναφοράς δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να είναι διάφανη όταν υπάρχουν ε, ε, παραπομπές κρατών μελών διότι υπάρχουν μεν συγκαλύψεις αλλά δεν είναι δυνατόν όλα να μένουν συγκεκαλυμμένα είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλεται η διαφάνεια και ίσως αυτό μπορεί να γίνει και μέσω των τροπολογιών και να αλλάξει κατά αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως δεν θα χρειαστεί να γίνει πολύ μακριά αυτή η οδός, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι κοινωνικές παροχές, ασυγχρόνως όμως και η συμμετοχή των πολιτών διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δούμε εάν είναι συνυπεύθυνοι οι οι πολίτες ε, και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαφάνεια και σε αυτό το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι ε, εγώ ε, ε, ζήτησα να δοθεί το έγγραφο αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας είπαν, μου είπαν ότι μπορείτε να το διαβάσετε αλλά πρόκειται για εμπιστευτικό έγγραφο άρα και οι πολίτες προσκρούν στο ίδιο θέμα και δεν είναι δυνατόν να τους λέει κανείς έτσι ψυχρά ότι δεν έχετε δικαίωμα να το ερευνήσετε Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει διαδικασία και κλεισμένων των θυρών διαφορετικά. Πρέπει ε, να υπάρχει διαφάνεια. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα το οποίο δεν βρίσκω αυτή τη στιγμή. Ε, και θα έπρεπε να τονίσουμε. Επίσης, αν ε, δω ότι βρίσκω αυτό το σημείο στο οποίο αναφερόμουν, θα επανέλθω αμέσως. Το βρήκα στην παράγραφο 4, ε, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 1049 του 2001. Ε, είναι το άρθρο 4 παράγραφος 2 λέει η κυρία Όκεν. Ευχαριστούμε την κυρία Όγκεν. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρτιν Κρόγκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, ζητώ συγγνώμη διότι είχαμε λίγη καθυστέρηση λόγω της αλλαγής ε, στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό που άκουσα ήταν το άκουσα της διαφάνειας. Θα ε, σχολιάσω γι' αυτό. Αν υπάρχουν και άλλα θέματα, αν θα μπορούσατε να υποβάλλετε ξανά την ερώτηση, την διευκρινήση που απαιτείται από την Κομισιόν. Για το θέμα της διαφάνειας γνωρίζετε ότι η Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο έχουν συμφωνήσει στο νέο πλαίσιο, συμφωνία πλαίσιο που περιλαμβάνει συγκεκριμένη διάταξη για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αρχεία παράβασης με δύο υποχρεώσεις ε, από πλευράς της Κομισιόν να παρέχει ε, συνοπτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις κατα... επί που τις παρέχουμε μέσα από μια ιστοθέση και ad hoc κατά ε, απέτηση παροχή πληροφοριών για τα ζητήματα που σχετίζονται με συγκεκριμένα υποθέσεις κατά παράβαση και έχουμε διευθετήσεις να παρέχουμε πληροφορίες στο Κοινοβούλιο σε αυτό το θέμα. Αυτή είναι η βάση που ακολουθούμε και ε, τα γενικά έγγραφα αναφοράς τα οποία θα ε, παρέχουμε ε, στο Κοινοβούλιο για πληροφορίε που αφορούν υποθέσει κατά παράβαση. Λοιπόν, αν ε, μπορείτε να μου ξαναποβάλλετε τις ερωτήσεις στα προηγούμενα ζητήματα, είμαι στη διάθεσή σας τώρα. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα. Μπορείτε... το μεγαλύτερο μέρος είναι η γνώμη μου. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν βρήκα αυτή την παράγραφο, διότι αυτή η παράγραφος 2 που λέει ότι οι θεσμοί θα ε, αρνούνται πρόσβαση στα έγγραφα όταν η αποκάλυψη υποσκάπτει την προστασία του. Λέει συγκεκριμένα πότε θα ε, κλείνει. Και υπάρχει και το εμπορικό ε, συμφέρον εκεί. Μετά, και είναι αυτό που χρησιμοποιείται συνήθω. οι δικαστικέ διαδικασίες και νομική συμβουλή. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο δικαστήριο όταν έχουμε υπόθεση επί παραβάση. Και τώρα ε, μπορεί μια μέρα στο μέλλον να υπάρξει ε, υπόθεση στο δικαστήριο. Αλλά εκεί μπορεί να, μπορεί να κλείσουν όλα μπορούμε να πούμε ότι αυτό μπορεί να είναι ε, υπόθεση στο δικαστήριο, αλλά δεν μπορούν οι πολίτες, οι ΜΚΟ να ε, δουλέψουν αυτό και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ιδιώτες και της ΜΚΟ να συμμετέχουν. Και είναι γι' αυτό που θα πρέπει να δούμε περισσότερο και να το συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το σημείο Ο Κρόγκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσα σας να κάνω μία απόπειρα να σας διευκρινίσω το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1049. Ως γνωρίζετε, ο κανονισμός 1049 αφορά αιτήματα για πληροφορίες και πρόσβαση σε έγγραφα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένο κανονισμός που να ρυθμίζει την πρόσβαση του Κοινοβουλίου σε ε, θέματα τα οποία ακολουθούν διαδικασία επιπαραβάση. Επομένως, αυτό το οποίο δίνεται στον κάθε πολίτη θα μπορούσε, και αυτό είναι λογικό, είναι τον Ονουκάνευ, να δίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, είναι λίγο πιο περίπλοκο το πράγμα, διότι υπάρχει νομολογία από το δικαστήριο που λέει ότι κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας όταν κάτι εκκρεμεί, τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα σε εμπιστευτικότητα ε, στα έγγραφά τους ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα βρεθούν ιδέουσες λύσεις σε συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη νομολογία και γι' αυτό ακριβώς στον 1049 υπό ομαλά συνθήκας δεν μπορεί να δοθεί καμία πληροφορία σε ατομικά αιτήματα από ε, πολίτες. Ένα άλλο μέσο τώρα είναι η συμφωνία πλαίσιο η οποία πηγαίνει πέραν των δικαιωμάτων των πολιτών και έχουμε εκχώρηση ειδικών δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για διαδικασίες οι οποίες είναι εν εξελίξη. Και το πλαίσιο το οποίο το διέπει είναι η πρόσφατα υιοθετηθήσα συμφωνία πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλει κάποιος το λόγο από τους συναδέλφους, η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Ω κοιόδης εισηγήτρια, με συγχωρείτε, θα ήθελα να πω μερικά λόγια σχετικά με αυτή την ετήσια έκθεση που τονίζει τη σημασία της σωστής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορούν να διασφαλίζονται με καλύτερο τρόπο. Αυτή η έκθεση επίσης δείχνει ότι τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νομοθεσίας έχουν οριμάσει αυξάνουν την συνεισφορά τους στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παρακολούθησης. Όπως ε, ανάφερε και η κυρία Άουκεν στην έκθεσή της, τα προβλήματα μεταβίβασης των ε, οδηγιών αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή κοινοτική νομοθεσίας. Τα εργαλεία για να το αποφύγουμε αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν ως αποτέλεσμα. Ακόμη και οι περισσότερες αναφορές δεν αφορούν παραβάσεις, παρέχουν στο Κοινοβούλιο και την Κομισιόν σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμες πληροφορίε για τις ανησυχίες των πολιτών. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω μια άλλη σημαντική πτυχή από την έκθεση της Κομισιόν μπορεί να αναφερθεί ότι η ε, προστασία του περιβάλλοντος ή θέματα εσωτερικής αγοράς συνεχίζουν να αποτελούν θέμα ενδιαφέροντος των περισσότερων αναφορών. Ε, περίπου 173 αναφορές, από τις οποίες 83 είναι καινούριε. Για να συνοψίσω, χαιρετίζω την πρόσκληση της Κομισιόν προς τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν ενεργά στον εντοπισμό ε, και την ανάληψη μέτρων, ε, προληπτικών μέτρων για κάθε νέα ε, νομοθετική πράξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μπασέσκου. Άλλες παρεμβάσεις. Απαντήσεις από πλευρά της κυρία Σόκεν. Really because... Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήμουν αρκετά καλή και θα έπρεπε να το παραδέχομαι όταν κάνω λάθος. Θα ήθελα να προσθέσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η παράγραφος που σας ανέφερα και νομίζω ότι και το δικαστήριο θα το υποστηρίζω, λέει ότι αν δεν υπάρχει ε, δημόσιο συμφέρον προς την αποκάλυψη των πληροφοριών. Θεωρώ αυτό είναι, ότι αυτή είναι η βασική αρχή που αφορά τη διαφάνεια. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συνολική παρέκκληση για τη διαφάνεια αυτή. Νομίζω ότι είστε πολύ νότιος και τα κλείνετε όλα. Είναι πολύ πιο εύκολα να είναι κλειστά τα πράγματα και πιστευτικά, το γνωρίζω, αλλά υπάρχει μια συνεχιζόμενη μάχη για να έχουμε διαφάνεια και νομίζω ότι υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου που το υποστηρίζει, αλλά θα το εξετάσω, να το εξετάσουμε και όλοι μας. Είμαι βέβαιη όμως ότι δεν είναι τόσο απλό όσο μας λέτε. Ευχαριστούμε κυρία Όκεν. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι Έχουμε προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για τις 2 Μαΐου για τη γνωμοδότηση στις 6 το απόγευμα και η γνωμοδότηση θα ψηφιστεί στην ε, ε, συνεδρίαση της 24ης Μαΐου. Εάν λοιπόν ο συνάδελφος Τσίτσεστερ συμφωνεί, θα ήθελα τώρα να του δώσουμε το λόγο γιατί συζητήσαμε πρώτα το σημείο 9 για τη γνωμοδότηση της κυρίας Άουκεν επειδή απουσιάζεται. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Τσίτσεστερ τώρα. Thank you, Chairman. Uh, uh, Ευχαριστώ πρόεδρε και λυπάμαι. Με συγχωρείτε για αυτή την uh, απουσία. Έχω την τιμή να παρουσιάσω αυτή το σχέδιο γνωμοδότησης στην Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία για τη βοήθειά της στη σύνταξη αυτού του σχεδίου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι προσπαθούμε να δούμε ορισμένα παραδείγματα υποθέσεων που έχουν ε, υποβληθεί σε αυτή την Επιτροπή που δείχνουν ότι είναι συναφή ε, και με ναι, θέματα ε, της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης ε, σχετικά με την κινητικότητα και την ενσωμάτωση ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και υπάρχουν πολλά, πολλά παραδείγματα και τα έχουμε δει μέσα από αναφορές. Δεν νομίζω να πρέπει να πω πολλά περισσότερα στο θέμα αυτό, απλά να πω ότι φυσικά καλωσορίζω τα σχόλια των συναδέλφων στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προσθέσουμε κάτι ή να ε, επιφέρουμε τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, ο κύριος Γκρέκο. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τσίτσεστερ για τις εισηγήσεις σας ε, στη γνωμοδότηση του κυρίου Κώσου. Καλωσορίζουμε αυτές τις εισηγήσεις και θα μπορούσα να κάνω κάποια σχόλια για μερικές. Δεν θα επισέλθω σε όλες τις λεπτομέρειες, εκτός αν ε, μου ζητηθεί συγκεκριμένα από τη δική σας πλευρά. Γνωρίζουμε, επειδή συμμετέχουμε στην, ε, σε τη της Επιτροπής Αναφορών. Ε, λαμβάνουμε και εμείς ε, τις αναφορές που υποβάλλονται εδώ και γνωρίζουμε, γνωρίζουμε ποια είναι τα κυριότερα θέματα αυτών των αναφορών. Τα περισσότερα σχετίζονται με θέματα που δεν είναι ευρωπαϊκής, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά όμως ορισμένα είναι πολύ συναφή για μας. Πρώτα απ' όλα, στο θέμα της προστασίας κατά των διακρίσεων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία κατά των διακρίσεων, Τώρα είναι περιορισμένο στους τομείς απασχόλησης, επαγγελματική κατάρτισης. Υπάρχει η οδηγία 2070-78. Υπάρχει μια πρόταση ή οδηγία που ενέκρινε ε, η Επιτροπή τον Ιούλιο του 2008 στην επέκταση σε άλλα θέματα πέραν της απασχόλησης, πρόσβαση στην παιδεία, πρόσβαση στα αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό, κοινωνική προστασία κλπ. Όπως θα γνωρίζετε, αυτή η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση στο Συμβούλιο γιατί στηρίζεται στο άρθρο 19 της συνθήκης και γίνεται ακόμη συζήτηση στο θέμα αυτό και βλέπω ότι μια εισήγηση είναι προέκταση του πλαισίου προστασίας κατά των διακρίσεων στο ε, με βάση τις ε, αναπηρίες. Ε, γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να έχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο επί του θέματος. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά την προσπελασιμότητα, την βελτίωση της πρόσβασης στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στις πληροφορίες και τεχνολογίες πληροφορικής είναι μία από τις κυριότερες δράσεις, τις οποίες ανακοίνωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωση Νοεμβρίου 2010 για τη στρατηγική, Ευρωπαϊκή, ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αναπηρίας 2010-2020. Τώρα προετοιμαζόμαστε προς ε, μια ε, ενδυνάμει πράξη, ευρωπαϊκή πράξη για θέματα αναπηρίας, ε, δηλαδή μέτρα βελτίωσης της προσπελασιμότητας, της πρόσβασης. Βέβαια το χρονοδιάγραμμα δεν έχει προσδιοριστεί, είναι ακόμη πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα, πρέπει να συζητηθεί με κράτη-μέλη, σε πρώτο στάδιο έχουμε και τους ενδιαφερόμενους και τους συμμετόχους, τους προσώπους των επιχειρήσεων, των οργανώσεων ε, αναπήρων. Ε, είναι πολλοί συμμέτοχοι που έχουν το λόγο σε αυτό το θέμα. Αλλά μέχρι τον επόμενο χρόνο η Επιτροπή θα δει κατά πόσο μπορεί να έχει μια πρόταση για ε, αυτή την πράξη, ευρωπαϊκή πράξη στα θέματα αναπηρίας με σκοπό τη βελτίωση της προσπελασιμότητας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες. Τώρα, στο σημείο 8 αναφερθήκατε στη χρήση της ε, κάρτας στάθμευσης, Ευρωπαϊκής Κάρτας Στάθμευσης Αναπήρων. Είναι πολύ καλό παράδειγμα ε, προώθησης της ε, κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άτομα με αναπηρίες είναι η σύσταση 1998 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εισήγαγε αυτή την μπλε Κονκάρτα, ε, το μοντέλο ε, που χρησιμοποιούν ε, άτομα με αναπηρίες για στάθμευση και αναγνωρίζεται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη τώρα. Τώρα, στην προέκταση αυτής της αμοιβαίας αναγνώρισης ωφελημάτων και δικαιωμάτων αναφέρατε την εισαγωγή μιας κοινή κάρτας ταυτότητας ατόμων με αναπηρίες. Βέβαια αυτό είναι πολύ πιο περίπλοκο το θέμα με την ανακοίνωση για την στρατηγική αναπηρίας που θα εγκριθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, η Κομισιόν λέει ότι θα ε, μελετήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ένα δίκτυο ακαδημαϊκών εμπειρογνωμών σε θέματα αναπηρίας από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία μελετούν αυτή τη στιγμή ε, αυτές τις επιπτώσεις ε, επί ε, αυτών των ευρημάτων θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορώ να σας πω περισσότερα για αυτό το θέμα, αλλά είναι βέβαια ένα πολύ σημαντικό σημείο της στρατηγικής μας. Το τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω αφορά το σημείο 11, ανάγκη για άτομα ε, με αναπηρές να έχουν αποτελεσματική ε, κοινωνική προστασία και μείωση της φτώχειας. Βέβαια υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι μια από τις εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει και το θέμα ε, της αναπηρίας. Είναι ένα κύριο ζήτημα και περιλαμβάνεται λοιπόν σε αυτή την ε, πλατφόρμα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Όκεν. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Σκιώδης χρειάστηκε να φύγει και θα κάνω μία παρατήρηση. Όπως ε, ανέφερε στην ε, μη ε, στην έλλειψη διακρίσεων πρέπει να μην υπάρχουν διακρίσεις κατά των κινητικά ε, ε, των ατόμων με ε, ειδικέ ανάγκες. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται από πλευράς αρχών, γιατί ήμουν στο Δανικό Κοινοβούλιο επί σειρά ετών, εγκαταστήσαμε πολύ δαπανηρά σανσέρ και έπρεπε όμως να το πράξουμε και αυτό που κάναμε ήταν ε, ώστε να μπορούν ε, να τα χρησιμοποιούν οι, ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Άρα το affordable πρέπει να έχει διπλή σημασία, δηλαδή και να διατίθενται και να μπορούν να τα καλύψουν. Ευχαριστώ. Άλλες παρατηρήσεις, ο κύριος Τσίτσεστερ θέλει κάτι να προσθέσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς αυτό είναι ένα ευχολόγιο. Και αυτά που είπε η κυρία Όκεν τα σημείωσα σχετικά με τη χρήση του όρου affordable, δηλαδή ε, που, γιατί και εγώ το διατυπώνω με την πλέον ευρεία σημασία του όρου ε, εάν τα άτομα μπορούν ε, να ε, πληρώσουν κάτι ή εάν κάποιος πρέπει να μπορέσει να καλύψει το κόστος αυτό. Και γενικώ ο όρος affordable έχει διάφορες σημασίες. Αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι από εμά είναι πολύ τυχεροί διότι δεν αντιλαμβάνονται πόσο δύσκολη είναι η ζωή των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Ορισμένοι βλέπουν τις επιπτώσεις. Όταν πάμε εις, στα σανσέρ εδώ, ε, εγώ είμαι ψηλός και ε, μειώνεται η όρασή μου γιατί γερνάω και πρέπει να σκύψω για να δω που είναι το σωστό κουμπί. Σκεφτείτε τι γίνεται αντιστρόφως με τους ανθρώπους που είναι σε αναπηρικές καρέκλες. Και ε, ε, ε, αν εγώ σκύβω δεν έχει σχέση με τη δυσκολία που έχει το άτομο στην αναπηρική καρέκλα ιδίως αν δεν υπάρχει ένα σανσέρ. Άρα είναι θέματα που πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα επιλύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω ότι και για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 4 Μαΐου στις 6 το απόγευμα και το έγγραφο θα ψηφιστεί στην ε, συνεδρίαση της 24 Μαΐου. Να περάσουμε τώρα τις ε, τρεις αναφορές που είναι γεγραμμένες στο σημείο υπαριθμών 12 της ημερήσιας διάταξης, η 11-10 του 2008 της Μέρι Ολύρη, η 12-96 του 2008 της Τζοζεφίν Μέρι Μάκεϊ και τις 10-37-2010 της Σέιμι Κάλεν. Είναι παρούσες οι αναφέρουσες. Είναι παρούσα, συγγνώμη, η κυρία Μέρι Ολύρη, στην οποία δίνω και απευθείας το λόγο. Παρακαλώ. Madam Κυρία Πρόεδρε, θέλετε να διαβάσω την αναφορά μου. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφερών που ενδιαφέρθηκε για την υπόθεση αυτή και μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω και να εκπροσωπήσω την κοινότητά μου εδώ. Θα ήθελα να σα μιλήσω για το θέμα των τοξικών αποβλήτων που βρίσκονται στο νησί του ε, Κόρκ ε, στην Ιρλανδία. Υπέβαλα στην αναφορά κάποια στοιχεία, μπορείτε να τα έχετε και εδώ εφιστώ την προσοχή σας σε κάποια θέματα. Το Κόρκ είναι ένα από τα μεγαλύτερους και πιο θεματικούς φυσικούς οικοτόπους. Είναι ένα πολύ ωραίο λιμάνι με φυσικές και... Ε, προστατευμένες περιοχές και βρίσκονται όλα στο κέντρο του νησιού. Υπάρχει λοιπόν ε, ένας ε, χιτά τοξικών αποβλήτων εκεί και ανησυχούμε για το γεγονός ότι δεν αναλαμβάνεται δράσεις Έχουν ε, υπάρξει πολλέ εκθέσει τα τελευταία 16 χρόνια, αλλά δεν έχει αναλυφθεί καμία δράση. Όλε οι εκθέσει από το 1998 μιλάνε για την ε, επιμόλυνση του λιμανιού από το ε, χιτά που υπάρχει εκεί και υπάρχει και ε, διαρροή σε πολλές περιπτώσεις. Στην έκθεση του 1996 δεν υπήρχε κανένας κανονισμός, ε, υπήρχαν 100.000 τόνοι ε, από τη Χαλιβουργία ε, τότε και θεωρούμε ότι δεν έχει ρυθμιστεί η κατάσταση από το 1996. Οι κυβερνητικές αρχές ανέλαβαν την ευθύνη το 2001 και η Chase ισχυρίζεται ότι βάσει της πράξης διαχείρισης αποβλήτων του 2005 η πράξη 75442 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ε, που είναι οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν έχουν καταφέρει να διαχειριστούν καταλήλως τα απόβλητα. Όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλη μόλυνση έχει υπάρξει τα τελευταία 16 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα και στο, ε, λιμάνι του Χάρμπορ δεν έχουν γίνει όσα πρέπει. Του Κόρκ, συγγνώμη. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την προστασία τη δική μας και για το περιβάλλον μας. Δεν ε, έχει ληφθεί κανένα μέτρο, οι ρυθμιστικές αρχές δεν δίνουν τη δέουσα προστασία και γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ εγώ σήμερα. Μία πρόσφατη έκθεση λέει ότι το λιμάνι του Χάρβορτ έχει ε, από τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνο στην Ιρλανδία, 44% άνω του μέσου όρου και είχαμε και μία ε, μελέτη 13 ετών που λέει ότι οι πάσχοντες στο ΚΟΡΚ έχουν ένα ανεξήγητο καρκίνο των όρχεων με ένα ποσοστό 27% ανώτερο του μέσου όρου σε εθνικό επίπεδο. Επομένως τα όσα συμβαίνουν δεν είναι δίκαια. Δεν έχει γίνει καμία πρόσφατη μελέτη για την περιοχή του λιμανιού, παρά το γεγονός ότι οι τοπικές αρχές ε, και από εκθέσεις υγείας της κυβέρνησης ε, έχουν ζητηθεί αντίστοιχες μελέτες, φαίνεται ότι κανείς δεν ε, ασχολείται με την υγεία της. Θα πρέπει λοιπόν τα συστήματα να λειτουργούν αποτελεσματικά και θα πρέπει να το ζητούν αυτό οι ευρωπαϊκές κοινότητες και θα πρέπει επίσης να πληρούν και το ρυθμιστικό τους ρόλο ε, δόθηκε και μια νέα έκθεση το 2008 και παρά το γεγονός ότι καμία από τις προηγούμενες συστάσεις και τις προηγούμενες εκθέσεις ε, που έχουν ζητηθεί από την κυβέρνηση δεν εφαρμόστηκαν. Η έκθεση του 2008 δεν ενθάρρυνε και ανέφερε ε, κάποιες βασικές περιοχές ανησυχίας. Υπάρχουν ε, πολύ ψηλά κατόφλια για τα ε, βιομηχανικά απόβλητα, ενώ κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται τα κατώτερα όρια για, τα, ε, ε, για την περίπτωση που έχουμε κατοίκου κατοίκους στις περιοχές. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται επίσης και με την επίδραση της σκόνης και με την επιμόλυνση στην διατροφική αλυσίδα. Όλα αυτά τα θέματα με ανησυχούν. Το Κόρκ βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και ε, η έκθεση δεν αντιμετωπίζει την πραγματική κατάσταση και τα συμπεράσματα που δίνει είναι παραπλανητικά. Το δεύτερο σημείο που μας ανησυχεί στην έκθεση είναι ότι η Young White Green ε, α, έδωσε ένα σημαντικό ποσοστό συγκέντρωση τοξικών ουσιών που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν από την Γεωτεχνική Έκθεση του 2005 και οι τοξικές ουσίες που δίνονται είναι, ε, εξα, αναφέροντας την έκθεση του 2005, ε, από κάποιο θαύμα εξαφανίστηκαν. Δεν τις διαπιστώνουμε πουθενά. Έχουμε μια εξέταση το 2009 και εκεί έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά τοξικότητας, ε, κυρίως ε, στο δείγμα 1 εδάφους. Τα δείγματα δείχνουν ότι υπάρχει επιμόλυση από βαρέα μέταλλα από το Holbau Online Site. Τώρα, το τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουν γίνει διάφορες συστάσεις τα τελευταία χρόνια για το πώς μπορεί να ελεγχιστοποιηθεί η ρήπανση. Η άδεια που δόθηκε από το EPA το 2001 λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό τείχος ε, γύρω από τις επιμολυσμένες περιοχές αλλά δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Η οδηγία 2006 κάθετος 12 στο άρθρο 6 ζητά να υπάρχουν σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για να μπορέσουμε να ε, διαθέσουμε επικίνδυνες ουσίες δεν είναι δυνατό να αφήσουμε ένα μολυσμένο χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε να ελέγξουμε τη μόλυνση. Όπως το ποσοστό της μόλυνσης είναι πολύ σοβαρό και σε πολλές εξαίσεις που έχουν γίνει υπάρχουν στοιχεία. Υπήρχαν 10 χρόνια ευημερία όπου υπήρχαν κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα και ωστόσο δεν έγινε τίποτα. Η κοινότητα φοβάται ότι θα ξαναμπεί ε, στο χρονοτούλαπο η όλη αυτή η ιστορία και δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το ζήτημα. Υπάρχει μόλυνση στο λιμάνι του Κόρκ, υπάρχουν και υψηλά κύματα, υπάρχουν και χώροι οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι και ε, λόγω του ξηρού καιρού δεν έχει γίνει τίποτα δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Τα τελευταία 16 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Η κοινότητά μας έκανε πολλά για να μπορέσουν να μας λάβουν σοβαρά υπόψη. Δυστυχώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε η Επιτροπή σα να ε, εξετάσει την αποτυχία των Ιρλανδικών αρχών να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και να μας βοηθήσετε να ακολουθήσουμε όλου του κατάλληλου διάβλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Äh, Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, καταρχήν ε, ε, με συγχωρείτε η κυρία Ματσόνη χρειάστηκε να αποχωρήσει για μία συνέντευξη τύπου και μετά θα επανέλθει εγκαίρως πριν φτάσουμε στους συντονιστές. Τώρα έχουμε συνοψίσει τρεις αναφορές στο σημείο 12 και τώρα έχουμε ε, την ε, ε ήταν η 11-10 2008 το 12-96 του 2008 και η 10-37 του 2010 Έμι Κάλεν ή της κυρίας μακέι και τα τρία θέματα αναφέρονται στο ίδιο σημείο και ουσιαστικά Ε, με προσκάλεσε ο τοπικός πληθυσμός και τρόμαξα διότι είδα ότι είχαν 37% περισσότερους καρκίνους από ό,τι η υπόλοιπη χώρα. Άρα ο τοξικός αυτός ο χώρος διέρε ε, αέρια ε, και ε, επηρέαζε την υγεία των κατοίκων ιδιαιτέρως όταν ε, διαπίστωσα ότι το 2005 διαπιστώθηκε σαφώς ότι αυτό δεν ε, συνάδε την νομοθεσία η οποία έλεγε ότι όλοι οι τόποι υγειονομικής ταφής έπρεπε να, να, ε, να έχουν μία άδεια και αυτό δεν συνέβαινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπάρχουν τρία βασικά θέματα και το πιο προφανές και το πιο ανησυχητικό είναι αυτό της ανθρώπινης υγείας διότι οι άνθρωποι είναι βασικό μέλημά μας για να μπορεί λοιπόν να συνεχίσει να λειτουργεί αυτός ο χώρος χωρίς ε, να γίνει μία μελέτη της υγείας ε, του πληθυσμού και να δούμε τι σχέση έχει ε, η ύπαρξη ενός τοξικού χώρου υγειονομικής ταφής με την κατάσταση των ε, ατόμων που κατοικούν σε αυτή την περιοχή ήταν μεγάλη αμέλεια και ε, ε, εσείς ασχολείστε εδώ με περιβαλλοντολογικά θέματα. Επίσης από πλευράς τουριστικής εξαρτώμαστε ή μιλάμε για μια περιοχή η οποία εξαρτάται από τον τουρισμό και άρα αφενός είναι πάρα πολύ άσχημο ο χώρος αυτός έτσι όπως παρουσιάζεται και ε, έρχονται ένα σωρό επιβατικά τα οποία φτάνουν στο λιμάνι του Κόρκ και ε, αντιμετωπίζουν αυτό το έσχος που επηρεάζει πολύ δυσμενώς τον τουρισμό και δεν βοηθά κανένα μας. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ετήσεως της Επιτροπής Αναφορών να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει, να αποφασίσει ποιος είναι υπεύθυνο, ποιος ευθύνεται γιατί α, γυρίζουμε γύρω γύρω εδώ και 10 χρόνια. Ε, πρέπει λοιπόν να πούμε ποιος ευθύνεται, να γίνει μία μελέτη η οποία να αποδείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του χώρου και των περιστατικών καρκίνου και τρίτον να κλείσει αυτός ο χώρος και να καθαρίσει και δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Αναφορών για να γίνει κάτι το οποίο ορισμένοι θεωρούν σαν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ακούσατε τις συναδέλφους μου εδώ και ε, τώρα η άλλη συνάδελφος η Όλα θα ε, μας πει επίσης τη δικιά της άποψη. Όλα Μακάρθη από το Εθνικό Μητέα του Κόρκ. Χαίρομαι που αντιπροσωπεύω την μελέτη εδώ εκ μέρου ε, τη Amy Collin, που είναι η πρόεδρο. Θέλαμε να υποβάλουμε αναφορά στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με τι ανησυχίε στα θέματα υγεία και περιβάλλοντο στο Hobble Island. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ευρωβουλευτή Σον Κέλλιν που υπέβαλε αυτή την ε, αναφορά εδώ. Το Hobble είναι ένα νησί που έχει μια ναυτική βάση στο Κόρκ. Ε, το κοβάλεντ είναι ακριβώς απέναντι. Το κόρκ είναι ε, μια μαύρη κοιλίδα για τον καρκίνο στην Ιρλανδία και πιστεύουμε ότι μια περιεκτική μελέτη υγείας θα πρέπει να εκπονηθεί για να αποδειχθεί ή όχι ο συσχετισμός με τα τοξικά απόβλητα που απορρίπτονται εκεί. Ο προηγούμενο ε, Υπουργό Περιβάλλοντο είχε υποσχεθεί τη δεξαγωγή μια μελέτη, αλλά αυτό δεν έγινε το 2010. Η προηγούμενη κυβέρνηση δαπάνησε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στο θέμα του Χολμπόλεν. Το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει πού δαπανήθηκαν αυτά τα χρήματα και για ποιου σκοπούς. Η χαλιβουργία ξεκίνησε να λειτουργεί στο κολμπόλον στι αρχέ του 50 και ε, περατώθηκε το 2001. Σχετικά με τα, τις ε, τοξικές το χρώμιο 6 έχει ε, εντοπιστεί. Αυτή η τοξίνη ε, έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρκίνο. Η τελευταία ανεξάρτητη μελέτη που έγινε από του White Green Young το 2008 συμπέρνε ότι το χρώμιο 6 και άλλε τοξικέ ουσίε μπορούν να μπαίνουν σε ρηχά και τα αποτελέσματα παρακολούθησης του αέρα έδειξαν ψηλά αποτελέσματα σε καιρούς ξηρού ε, κλίματος. Όπως ακούσατε και από τους προηγούμενους, το ποσοστό είναι 37% άνω του, μέσου όρου, του εθνικού μέσου όρου στην Ιρλανδία και είναι πολύ ανησυχητικό. Σχετικά με την αδειοδότηση, ε, το Συμβούλιο του ΚΟΡΚ είναι η αρχή διαχείρισης του λιμένα και είναι δική τους ευθύνη να εφαρμόσουν, ε, να ζητήσουν μια άδεια. Από τότε δεν έχουν αιτηθεί για άδεια. Γι' αυτό ε, τα απόβλητα βρίσκονται εκεί παράνομα. Δεν έχει ληφθεί καμία δράση από το Συμβούλιο του ΚΟΡΚ, της Κομιτέας του ΚΟΡΚ, παρόλο που η Κομισιόν έστειλε προειδοποιητική επιστολή για το καθαρισμό του χώρου. Σχετικά με το, την εντολή του Γραφείου Δημοσίων Έργων, αυτό το Υπουργείο, το Γραφείο θεσπίστηκε για να εξετάσει το θέμα. Η εντολή δεν εξετάζει τον περιορισμό του χώρου ή την επιμόλυνση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ασχοληθεί με την επιμόλυνση του χώρου και όχι την μελλοντική χρήση του χώρου. Οι τοξίνες ε, ε, επηρεάζουν ε, την ζωή στο λιμάνι του Κόρκ και μπορεί να σχετίζονται με τα ποσοστά και την επίπτωση καρκίνου στο Κόρκ. Θα πρέπει να ληφθούν επίγοντα στα βήματα για την αντιμετώπιση αυτών των τοξινών από το χρόνιο έξω. Συμπερισματικά υπήρχε ένας χώρος χειρονομικής ταφής τοξικών αποβλήτων στην περιοχή. Το Κόρκ δεν μπορεί να, να προσδιορίσει τι ποσότητες υπήρχαν. Οι πολίτες του Κόρκ αξίζουν ε, να έχουν μια καθαρή πόλη, ένα καθαρό χώρο. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια μελέτη και ζητάμε από αυτή την Επιτροπή να παροτρύνει ε, μια ε, περιβαλλοντικά ασφαλή περιοχή προς όφελος της προστασίας περιβαλλοντος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ντέβιτ Στάντον που τόνισε αυτό το θέμα για πολλά χρόνια σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και πάλι τον Σον Κέλλη, ο οποίος υπέβαλε αυτό το θέμα σε, ε, στο επίπεδο του, της Επιτροπής αυτής. Σας ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ τους αναφέροντες και τώρα έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τοποθετηθεί. Ο κύριος Πρέκλεντ. Σωστά ε, παρουσίασα το όνομά σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι από πλευρά γεγονότων συμφωνούμε απολύτω με του αναφέροντες. Η κατάσταση επιτόπου είναι επικίνδυνη και πολύ ε, περίπλοκη. Υπάρχει ένα τοξικό ναρκοπαίδιο χωρίς καμία άδεια. Γι' αυτό και ακριβώς ε, ξεκινήσαμε ε, κατά της ε, Ιρλανδίας διαδικασία. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ιρλανδία για συστηματική αποτυχία να διαχειριστεί καταλήλως αυτούς τους χώρους υγειονομικής ταφής και συγκεκριμένα τους συγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ζητήσει να πιέσουμε την Ιρλανδία και... Έχουμε στείλει και συγκεκριμένη επίσημη κοινοποίηση βάσει του άρθρου 260 της συνθήκης και έχουμε επιβολή προστήμων για να τηρήσει η Ιρλανδία τις υποχρεώσεις της και ζητείται να καθαριστεί ο χώρος και να μην ε, πάψει να υπάρχει ρήπανση. Σε προσωπική ε, σε προσωπικό επίπεδο να σας πω ότι και εγώ είμαι απογοητευμένος λόγω της καθυστέρησης των Ιρλανδικών αρχών ε, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Ξέρω ότι είχαμε υποσχέσεις στο παρελθόν, δεν τηρήθηκαν και πρέπει να πω ότι δόθηκε εντύπωση ότι ο νέος Υπουργός ε, Περιβάλλοντος είχε καταλάβει ε, πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσες προκλήσεις υπάρχουν για την ε, εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων στην Ιρλανδία και βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια κίνηση και σε άλλα θέματα. Λάβαμε ενημέρωση από τις Ιρλανδικές Αρχές ότι θα αναθέσουν την αρμόδια αρχή για τον καθαρισμό του χώρου εντός του μηνός αυτού. Θα δούμε βέβαια αν τα πράγματα πάνε καλά, μπορεί να έχουμε και καλά νέα να ανακοινώσουμε για τον καθαρισμό του χώρου. Αυτό είναι άλλωστε αυτό που επιθυμούμε. Αν όχι, εάν δεν υπάρχει ε, γρήγορα δράση από τις ελληνικές αρχές, θα ξεκινήσουμε ή τουλάχιστον ο Επίτροπός μου θα προτείνει να ε, περάσουμε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να προτείνουμε να επιβληθούν πρόστιμα. Όπως ε, γνωρίζετε προσφάτως ε, λάβαμε δράση κατά της Ιρλανδίας ήδη από το Φεβρουάριο και περιμένουμε πλέον αποτελέσματα από την ε, Ιρλανδία και για να πω αυτό που είπε και η κυρία Ολύρη δεν θα περιμένουμε άλλα δέκα χρόνια. Äh, Νομίζω ότι ήταν σαφής η απάντηση αλλά κάποιος έχει ένα σχόλιο. Ωραία. Μία απλή ερώτηση, ο κύριος Μασουνάρου, διότι είναι κάτι που διαπιστώνουμε καθημερινά. Πώς είναι δυνατόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επί 10 χρόνια να αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα σε ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν ήταν ένα νέο κράτος μέλος, θα, υπήρξε, θα υπήρχε κάποια απάντηση. Είναι λιγότερο καλά προετοιμασμένοι, λιγότερο εκπαιδευμένοι και μπορούσαμε να το δεχτούμε. Αλλά όταν μιλάμε για ένα παλιό κράτος μέλος, το οποίο ε, συνεχώς ε, και επισταμένος είναι σε τέτοια κραυγαλαία παραβίαση και ε, ε, ε, να συνεχίζει πιστεύω ότι πρέπει όχι μόνο να μας τρομάζει αλλά να θεωρήσουμε ότι είναι απαράδεκτο. Και αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι μία έκθεση για τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες και τους κανονισμούς. Γιατί είναι τόσο διστακτική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ζητά πολύ πιο αυστηρές ποινές και, και συνθήκες ώστε να ε, αποκαταστήσει το πρόβλημα όταν εμφανίζεται σε τέτοια έκταση διότι αφενός καταστρέφουμε το περιβάλλον και από την άλλη πλευρά καταστρέφουμε μέχρι και την βιοπικιλότητα. Τώρα διαπραγματευόμαστε με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και προσπαθούμε να τους διδάξουμε, να τους πούμε τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να βελτιωθεί, τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσμονές μας. Και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα τόσο κραυγαλαίο παράδειγμα και δεν είναι και το πρώτο. Διότι η περίπτωση της Ιρλανδίας δεν ξέρω πόσες άλλες τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν με ακριβώς τα ίδια περιστατικά. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν. Και με την έκθεση αυτή και με τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν το φθινόπερο και πάλι κάνουμε μία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία πρέπει να μας προσεγγίσει, να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα διότι διαφορετικά το να λέμε ότι ε, είναι καλή και αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν μπορεί να ε, λύσει ε, μικροπροβλήματα δεν μιλάμε εδώ για μια παγκόσμια κρίση δεν μιλάμε για κατάρρευση της χρηματαγοράς ή της παγκοσμίου οικονομίας μιλάμε για ε, μία έκταση όπου ε, όλο η κατοικημένη περιοχή επηρεάζεται από την κακή διαχείριση των αποβλήτων. Ε, αυτό είναι που μας ανησυχεί, αυτή η παθητικότητα αυτή η ανικανότητα να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια πιο ικανοποιητική απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι μας είπατε ότι υπήρξε κάποια απόφαση, επευλήθησαν κυρώσεις και παρόλα αυτά να μην μπορούμε να πείσουμε μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μετά από τόσα χρόνια, δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι, μια, είναι εις βάρος όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κυρία Όκεν, απλώς συμφώνησα με αυτά που υπόθηκαν. Δεν ήθελα το λόγο. Ε, Α, σας υποστηρίζω. Και οι αναφέρουσες μπορούν να δευτερολογήσουν. Θέλουν... Ε, ε, έχω όμως και εγώ μια ερώτηση πριν σας δώσω το λόγο αντιληφθήκατε ότι κάτι θα αλλάξει διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας άφησε να νοηθεί ότι τις επόμενες εβδομάδες ή ημέρες ε, κάτι θα συμβεί. Ίσως τα μεγάλα γεγονότα ε, ανακοινώνονται εκ των προτέρων και ελπίζω ότι όλα αυτά μπορούν να σας οδηγήσουν στο να αναλάβετε κάποια δράση. Ευτυχώς τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν και χαιρετίζω τις δηλώσεις της Κομισιόν ότι ο καινούριος Υπουργός, ο κ. Κόγκαν, θα ασχοληθεί με ε, το θέμα ως επίγον σε αντίθεση με τον προηγούμενο Υπουργό. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα θα είναι σημαντικό παρά να λέμε ότι ελπίζουμε θα αναλυθεί, ε, να αναλυφθεί δράση να δώσουμε κάποια προθεσμία, να θέσουμε μια προθεσμία. Διότι το το συντομότερο δυνατόν τι σημαίνει, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε έξι μήνες. Για τους πληγέντες και αυτούς που επηρεάζονται, ιδιαίτερα 37% επίπτωση ψηλότερη από τον ε, μέσο όρο στους καρκίνους, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται άμεσες απαντήσεις. Δεν μπορεί να περιμένουν άλλο. Περίμεναν τα τελευταία 10 χρόνια. Γι' αυτό θα θέλαμε από την Κομισιόν να μας πούν συγκεκριμένα τι σημαίνει το συντομότερο δυνατόν. Επόμενη, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τις υποδείξεις της Κομισιόν ότι θα διοριστούν οι αρχές που θα αναλάβουν τον καθαρισμό του χώρου διότι είναι επίγον το θέμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η κατάσταση, η ανθρώπινη υγεία είναι πρωτής της σημασίας και κάθε 11 μέρες ένα άτομο διαγνώσεται με, διαγνώσεται με καρκίνο. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ε, και προσβλέπουμε στον καθαρισμό του χώρου ως θέμα επίκουσης σημασία. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε ε, μέρους της ομάδας για την υγεία των ανθρώπων του ΚΟΡΚ. Και εγώ με τη σειρά μου χαίρομαι που άκουσα από την Κομισιόν ότι κάτι θα συμβεί. Δυστυχώς το ακούσαμε και το 2008. Και τελικά εκπονήθηκε άλλη μια έκθεση χωρίς δράση και δεν ξέρουμε πού δαπανήθηκαν τα 50 εκατομμύρια. Εάν ε, δαπανήθηκαν για να γίνει κάτι, για να σταματήσει η εκροή των τοξι... της τοξικής ηλίως, ε, γιατί κάθε φορά που έρχονται τα νερά μέσα ε, στο λιμάνι, έρχονται μαζί και όλες οι τοξικές ουσίες αν σταματήσει αυτό θα δώσει κάποιο θάρρος στους ανθρώπους του ΚΟΡΤ. Ε, ελπίζω να μην είναι απλά λόγια, ελπίζω να περάσουμε στις, στη δράση. Σύντομα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επειδή υπάρχει μια απόφαση του ΔΕΚ και υπάρχει καθαρή παράβαση οδηγιών. Τι είδους δράση μπορεί να αναμένει κανείς στο να αναγκάσουμε τις τοπικές αρχές να συμμορφωθούν λόγω του ανεύθυνου τρόπου με τον οποίο χειρίστηκαν το θέμα. Διότι πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια σαφή υπόδειξη ε, και δράση που πρέπει να αναμένουμε να αναλυθεί, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής. Η Επιτροπή απάντησε σαφώς ότι υπάρχει παραβίαση, υπάρχει καταδίκη, υπάρχει διαδικασία παραβίασης, υπάρχει η δέσμευση της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι κάτι θα κάνουν στο άμεσο μέλλον, εντός των επομένων εβδομάδων. Λοιπόν, ε, καταρχήν στηρίζουμε τις αναφέρουσες ότι δεν είναι ανεκτή αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, δηλαδή την ε, έκθεση την οποία συζητήσαμε, πολλές φορές βλέπουμε ότι διαπιστώνουμε μία κατάσταση και ε, δυστυχώς παραμένουμε με δεμένα χέρια και χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα και βλέπουμε ότι στο πινκ πονγκ μεταξύ Επιτροπής και εμπλεκομένου ε, κράτους το κράτος μένει, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και αυτό πρέπει να το τονίσουμε και στην έκθεσή μας. Να αφήσουμε λοιπόν την αναφορά αυτή ανοιχτή, να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει και κατά δεύτερον λόγο σαν επιτροπή να απευθύνουμε μία επιστολή στην Ιρλανδική κυβέρνηση και να του πούμε για μια ακόμη φορά ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση και πρέπει να, ε, να σταματήσει. Ε, θέλει κάποιος να κάνει μία τοποθέτηση ή μία γνωμοδότηση του θέματος. Νομίζω είναι εξαιρετική αυτή η ιδέα και θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε από την Κομισιόν ας πούμε, σε μια περίοδο τριών μηνών, σε ένα χρονικό διάστημα, να επανέλθουν με μια έκθεση προόδου. Να μην το αφήσουμε έτσι ανοιχτό το θέμα, δηλαδή. Οι αναφέροντες θα έχουν μια σαφέστερη ιδέα για το πότε να αναμένεται αυτή η έκθεση προόδου. Γιατί αλλιώς μπορεί να παραμείνει εκεί, είναι μια επιτροπή με πολύ ε, πολλή δουλειά, με πολλές αναφορές, αλλά αυτή η ιδέα σας ήταν εξαιρετική. Σας ευχαριστώ. Απευθύνω και πάλι την ερώτησή μου στην Επιτροπή, η οποία ήταν ε, αισιόδοξη και μας είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες κάτι θα γίνει. Πότε ε, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας δώσει μία απάντηση για να προβλέψουμε μία προθεσμία στα πρακτικά διότι η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να υπάρξει επίλυση. Τρει μήνε νομίζω ότι είναι κατάλληλο χρονικό διάστημα. Ίσως έχουμε απάντηση και πιο πριν, αλλά πιστεύω εντός τριών μηνών είτε θα έχουμε καλά αποτελέσματα είτε θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες. Ευχαριστώ. Έχουμε και τον συνάδελφο Κέλλη. Κύριε Κέλλη, μπορείτε από καιρού καιρών να μας ενημερώνετε αν κάτι γίνεται ή όχι και σαν μέλη της Επιτροπής Αναφορών περιμένουμε να αναλυφθούν μέτρα και κάτι πρέπει να γίνει, κάτι ουσιαστικό εντός των επομένων εβδομάδων και ο κύριος Κέλλη παρακαλώ να μας ενημερώσει μόλις θα υπάρξουν εξελίξεις. Άρα μένει ανοιχτή η αναφορά. Δεύτερον, το πολύ σε τρεις μήνες θα επανέλθει και τρίτον θα απευθύνουμε μία επιστολή στην Ιρλανδική κυβέρνηση και να του ζητήσουμε επιγόντως και το ταχύτερο να καταργήσουν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση και εντωμεταξύ θα μας ενημερώνει για τα τεκτενόμενα ο κύριος Κέλλη. Ε, διότι εδώ διακυδεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όπως είπατε δεν πρόκειται για μία υποανάπτυξη χώρα, πρόκειται για μία ε, αναπτυγμένη χώρα κράτος μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, πρέπει απλώς να αποκατασταθεί η κατάσταση δικαίου. Κύριε Κέλ, μία τελευταία παρατήρηση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την κατανόησή σας και για την ε, πολύ ε, θετική σας αντιμετώπιση σήμερα και για τον τρόπο με τον οποίο συνοψίσατε με ικανοποιεί απολύτως. Επίσης ε, στην Επιτροπή θέλω να πω ότι τρεις μήνες προθεσμίας αρκεί και θα σας δοθεί ο χρόνος κάτι να γίνει και να δημιουργηθεί μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ότι εμείς ακούμε τους πολίτες και ε, αναλαμβάνουμε δράση μόλις ε, υπάρξει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και θα μείνει το θέμα ανοιχτό και εμεί θα μείνουμε με τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά για να σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Ευχαριστώ τις αναφέρουσες, ε, ε, τους, ευχαριστώ, τους εύχομαι καλό ταξίδι και ελπίζω να αποκομίσανε και μία θετική ε, εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 13 πάλι της Ιρλανδίας ε, που υπάρχουν τρεις ε, αναφορές 872, 883, 902 και 1207 τέσσερις. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Higgins θα μας διαβάσει μία δήλωση των αναφερόντων Εν ονόματι λοιπόν των αναφερόντων, πρόκειται να μιλήσετε πρώτος. Η κυρία πρώτη ή εσείς, ό,τι θέλετε, αποφασίστε μόνοι σας. Ε, θα τα πω εγώ. Καταρχάς, θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, ότι το Δεκέμβριο του 2009 έφερε εδώ τρεις οικογένειες, όπως έκανε και η κυρία Χάρκιν και ο κύριος Κέλλη, και όσον αφορά τις εξουσίες της Επιτροπής Αναφερών, να σας δώσω ε, το εξή παράδειγμα. Έχασαν τρεις όμορφες κόρες αυτές οι τρεις οικογένειες λόγω της αμέλειας των Ιρλανδικών αρχών. Αυτή την εβδομάδα όλες οι τοπικές αρχές κάνανε ε, ρυθμίσεις ε, με τις οικογένειες για αποζημιώσεις και αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή Αναφερών δεν είναι απλώς ε, ένα μέσο παραπόνων, έχει εξουσία. Η αριθμητική κυβέρνηση, οι τοπικές αρχές ε, αναγνωρίζουν ότι οι τρεις κοπέλες που χάθηκαν δεν ε, ήταν υπεύθυνε για το θάνατό τους και από πλευράς αποζημίωσης αναγνωρίζεται ότι οι Ιρλανδικές τοπικές αρχές ε, προτίμησαν να μην ε, εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές και έκαναν ε, ρυθμίσεις για αποζημίωση εκτός δικαστικής αιθούσης. Και αυτό δείχνει τι εξουσίες έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη υπόθεση την οποία παρουσιάζουμε εγώ και η κυρία Χάρκινγκ, αφορά τις πλημμύρες. Όταν υπάρχει μια πλημμύρα στην Ιρλανδία, δεν είναι σαν μια πλημμύρα στο Ρήνο που έχονται πλημμύρα τη μια μέρα και την άλλη μέρα έχουν εξαφανιστεί όλα τα νερά. Στη δική μας την περίπτωση, επειδή υπάρχει Υπάρχει ο σβεστόλαθος και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν μετά τις πλημμύρες προβλήματα τρει-τέσσερι μήνες μετά. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για κατοικίες που ε, καταστράφηκαν το Νοέμβριο του 2009. Οι οικογένειε αυτές έχασαν τα σπίτια τους. Ε, το νερά της πλημμύρας πέρασαν από την ε, πόρτα και μπήκαν στα σπίτια και καταστράφηκαν τα σπίτια του ολοσχερών. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να λάβουν αποζημίωση από την Ιρλανδική κυβέρνηση ε, και δεν μπορούν ταυτόχρονα να λάβουν και ασφαλιστική κάλυψη, διότι οι ιδιοκτησίες αυτές ε, βρίσκονται σε περιοχές ε, σχεδίων πλημμυρών. Το 1994 και το 1995 εγώ ήμουν υπουργό υπεύθυνο για τις πλημμύρε. και το 1994-1995 εγώ ζήτησα να εκπονηθεί μια μελέτη για το πώς ε, ε, θα ε, καθορίσουμε συγκεκριμένες περιοχές ευθύνη πλημμυρών και κάναμε μία χαρτογράφηση και στο χάρτη έλεγε ότι δεν θα πρέπει να δίνονται άδειες οικοδόμηση. Ε, ακόμα και σε γαστικά προγράμματα σε περιοχές που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χάρτη. Και στην περιφέρειά μου δόθηκαν πολλές ε, άδειες που είναι περιφέρεια και της κυρίας Χάρκινγκ στο κομιτεία του Κάλουεϊ να σας πω εδώ ότι μία από τις ε, περιπτώσεις έχει αποσυρθεί διότι ε, λόγω της απελπισίας τους η οικογένεια Μακάφ ε, μετανάστευσε στην Αυστραλία και δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Έχουμε λοιπόν τρεις οικογένειες εδώ. Την οικογένεια Κίναν, την οικογένεια Φλάτλη και την οικογένεια Κόνμποϊ. Και στις δύο περιπτώσεις που σας αναφέρω εδώ, στην οικογένεια Κίναν και Φλάτλη, δόθηκε άδεια ε, κατασκευής ε, άδεια οικοδομική, οικοδομική άδεια, σε μια περιοχή που εγώ έκανα μια έκθεση το 1994 και δημοσιεύτηκε το 1995 που έλεγε ότι απαγορεύεται να κατασκευαστούν κατοικίες εκεί, διότι υπάρχει ε, με πλημμύρες επαναλαμβανόμενο. Παρ' όλα αυτά δόθηκε οικοδομική άδεια και τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Οι οικογένειες αυτές δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν αποζημιώσεις και δεν έχουν δυνατότητα επανεγκατάστασης. Αυτό που έκανα εγώ το 1995 ήταν ε, να κάνω μετεγκατάσταση 400 ε, οικογενειών που ζούσαν εκεί. Δεν υπήρχε ασφάλιση, τους δόθηκε ένας νέος χώρος, δυνατότητα να κατασκευάσουν μια νέα κατοικία και ούτω καθεξής. Εάν δεν είχαν, ε, αν είχαν συγγνώμη κάλυψη, κάναμε μια εξωσυρήπηση με τη διαφορά. Δηλαδή τους δόθηκε ένα ποσό από την ασφάλεια και δώσαμε το υπόλοιπο εμείς. Η νέα κυβέρνηση που εξελέγει 25 Φεβρουαρίου του 2011 αρνήθηκαν να κάνουν το οτιδήποτε και δεν δίνει καμία αποζημίωση στις οικογένειες αυτές. Αυτό που σας λέω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση και δεν εξαρτώμεθα μόνο στην οδηγία για τις ε, πλημμύρες, διότι η οδηγία για ε, τις πλημμύρε θα βγει σε μερικούς μήνες. Μας ενδιαφέρουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και το τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτές τις οικογένειες. Οι οικογένειες που σας παρουσιάσαμε εμείς το 2009 δεν είχαν καμία ευρωπαϊκή οδηγία να τις προστατεύσει, αλλά λόγω των πιέσεων που δόθηκαν οι Ιρλανδικές αρχές ε, και ε, οι τοπικές αρχές ε, αναγκάστηκαν να ακουστεί η άποψή τους και τελικώς δόθηκε αποζημίωση για την απώλεια των τριών κοριτσιών. Και εμεί ζητάμε το ίδιο όριο ανοχής και κατανόησης σε αυτή την περίπτωση. Αυτές οι οικογένειες δεν έχουν σπίτια, οι κατοικίες τους καταστρέφηκαν επειδή κατασκευάστηκαν σε ε, περιοχές όπου απαγορευόταν. Ε, θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο και θα ε, δώσω το λόγο στην κυρία Χάρκιν. Πρόκειται για μια τοπική αρχή η οποία θα σας πει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη για τις πλημμύρες. Αλλά ταυτόχρονα θα σας πει ότι το χρώμα των κεραμιδιών που θα βάλετε στις σκεπή σα, το μέγεθος της πόρτας σας, το μέγεθος των παραθύρων σας, το μέγεθος της κατοικίας σας και η πρόσβαση σε ένα δημόσιο δρόμο είτε είναι ασφαλής είτε είναι μη ασφαλής, θα όλα καθορίζονται από εμά. Αλλά όταν πρόκειται για πλημμύρες μας λένε δεν έχουμε καμία σχέση, δηλώνουμε άγνοια. Στην ουσία κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι η αρχή και το τέλος ε, του επιχειρηματός μας. Η κυρία Χάρκιν. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι ο συνάδελφος έχει καλύψει τις λεπτομέρειες και πιστεύω το τελευταίο σημείο που έδειξε το έχει δείξει πολύ καλά. Εάν δεν σου αρέσουν ε, τα κεραμίδια, το έχεις πρόβλημα, αλλά δεν ασχολούνται καθόλου με το θέμα των πλημμυρών. Πιστεύω ότι το θέμα εδώ και η απάντηση από την Κομισιόν μας λέει, όπως γνωρίζαμε, ότι η ε, οδηγία περί πλημμυρών δεν είναι αδανδρομική. Θα να μιλήσω... Μιλάνε για την οδηγία περί ε, πτηνών και λένε ότι οι αναφέροντες δεν παρέχουν ε, περιστατωμένα στοιχεία επιστημονικά που θα πρέπει να ε, αποτελεί ζώνη δικής προστασίας. Αυτό είναι αδύνατον για έναν πολίτη να το κάνει, για έναν ιδιώτη να το κάνει, να παρέχει αυτές τις επιστημονικές, τα, επιστημονικά τεκμήρια και αποδείξεις που χρειάζεται χρόνια να τα συλλέξει κανείς. Για έναν ιδιώτη να πάρει μια τέτοια απάντηση, ακόμη και αν είναι επακριβής, δεν έχει κανένα νόημα και ε, δεν τους ενθαρρύνει. Ο κύριος Χίγκιν ε, εξήγησε την κατάσταση των ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Τώρα που έκτισαν τα σπίτια τους σε αυτή την περιοχή, δεν έχουν ασφάλεια, δεν υπάρχει σχέδιο αποζημίωση των πολιτών για αυτές τις καταστάσεις οι οποίες έχουν βρεθεί. Και αυτό που κάνουν, ε, ε, έχουν φέρει την υπόθεση εδώ στην Ευρώπη, παρόλο που δεν υπάρχει νομοθεσία που να την καλύπτει, αλλά όπως είπε, σε μια παρόμοια περίπτωση ε, κατάφεραν να βρουν επανόρθωση οι πολίτες και γι' αυτό αναφέρεται σε αυτήν την Επιτροπή, ακόμη και αν δεν έχει απόλυτη αρμοδιότητα μπορεί να έχει αντίκτυπο. Είναι ένα θετικό μήνυμα το οποίο πρέπει να ακούσουν όλα τα μέλη. Σας ευχαριστώ. Ποιος θα αναλάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Κασπαρανέτη. Ευχαριστώ και Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα έντιμα μέλη που ε, ήγηραν το θέμα. Η Επίτροπη γνωρίζει τα προβλήματα, παρόμοια προβλήματα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε τα έντυπα μέλη που έφυξαν το πρόβλημα της ανάγερσης οικειών στις περιοχές πλημμυρών. Είναι ένα πρόβλημα που αναφέρεται σε μια λευκή βίβλο για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, όπου λέμε ότι μεγάλες εκτάσεις, για παράδειγμα στο Λονδίνο, ε, μεγάλες οικιστικές ε, εκτάσεις που, είχαν άδειε χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ακραίες κλιματικές καταστάσεις μπορεί να είναι όλο ένα και πιο συχνές. Κατανοούμε ότι τα επεισόδια στα οποία αναφέρονται οι αναφέροντες ήταν ένα επεισόδιο ακραίου κλιματικού ε, επεισοδίου που συμβαίνει στην Ιρλανδία, αλλά με τις κλιματικές αλλαγές αυτά τα επεισόδια είναι όλα πιο συχνά παντού και όχι μόνο στην Ιρλανδία. Όπως ε, σωστά επέδειξε το έντιμο μέλος, ιδιαίτερα η, η, η, οδηγία για τις ε, πλημμύρες δεν έχει... δεν έχει ισχύ συνέχεια. Δεύτερον, εκεί που υπάρχει κίνδυνος μέχρι το 2013 θα πρέπει να ε, καταρτήσουν ε, χάρτες κινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας και μέχρι το 2015 τα σχέδια αυτά θα πρέπει να εκπονηθούν για τις ζώνες αυτές. Έχω συνοψίσει τις κύριες ε, προθεσμίες που έχει θέσει η οδηγία για τις πλημμύρες. Γι' αυτό είναι σωστό να πει κανεί ότι η οδηγία αυτή καθ' αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, διότι δεν έχει αναδρομική δράση ως βάση για αποζημίωση και αναφέρατε επίσης ότι ευρύτερα θέματα εδώ διακυβεύονται όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα για την δίκαιη αποζημίωση. Δυστυχώ δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά από πλευράς ε, κομισιών σε περιοχές που δεν είναι εναρμονισμένες και η, Κομισιόν κοιτάζει ε, υποθέσεις παραβάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου ε, συμπαραστεκόμαστε και θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάτι κάποιες τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν υπό το φως ε, της δικής μας εξέτασης των κλιματικών αλλαγών και του γεγονότος ότι αυτό θα συμβαίνει όλο ένα και πιο συχνά. Είχαμε πολλές υποθέσεις όπου το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, ε, χρησιμοποιήθηκε για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των πλημμυρών στην Ευρώπη. Είναι αυτό έχει συμβεί σε κάποια ε, κράτη-μέλη. Βέβαια, αν οι τοπικές αρχές ε, δίνουν άδειες οικοδομής σε περιοχές που έχουν εντοπιστεί, εντοπιστεί ως περιοχές πλημμυρών, είναι μια ε, περίπτωση που μπορούν να φέρουν ενώπιον του δικαστηρίου και ε, μέσα παρέχονται από το, τα εγχώρια δικαστήρια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ακόμη ένα σημείο. Θα πρέπει να αναφερθώ στο σημείο ε, σχετικά με την οδηγία για τα πτηνά. Έχει απόλυτο δίκιο η ε, ε, συνάδελφος και είναι δύσκολο βέβαια για ένα άτομο να παρέχει αυτές τις επιστημονικές πληροφορίες που ζητούνται. Από δική μας πλευρά έχουμε παρόμοιο πρόβλημα όμως το Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας έχει τις δικές του ε, εξουσίες ε, επιθεώρησης. Γι' αυτό και η συλλογή στοιχείων από τη δική μας, δικής μας είναι δύσκολη. Η Κομισιόν όμως πρέπει να έχει στοιχεία στη διάθεσή της ότι υπάρχει παραβίαση. Δεν θα σχολίαζα συγκεκριμένα αυτό το θέμα, αλλά είναι ένα γενικό πρόβλημα το οποίο ε, θα αναφέρουμε σε μια ανακοίνωση σχετικά με την βελτίωση αυτών των θυμάτων. Είναι σαφές όμως ότι ε, μπορούμε να βρούμε στοιχεία. Αν δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία δεν μπορούμε να ε, κάνουμε εμεί αυτέ τι επιθεωρήσει, άρα συμφωνώ με αυτό το θέμα, αλλά θέλω να κατανοήσετε ότι και η εξουσία τη Κομισιόν σε αυτό το τομέα είναι πολύ περιορισμένη. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, λοιπόν, τώρα τα μέλη τη Επιτροπής μπορούν και πάλι να παρέμβουν. Ο κύριο Κέλλη είναι ο πρώτο που ζήτησε το λόγο. Θέλω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους τον κύριο Χίγινγκς και την κυρία Χάρκινγκ και χαίρομαι και λυπάμαι διότι αφενός μπορούμε να ερχόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή αυτή και να μας ακούν. Και αυτό που με λυπεί είναι ότι και πάλι βλέπουμε ορισμένες από τις παρεκτροπές του κελτικού τίγλη και ε, ε, ε, μας επαναφέρουν στη θέση στην οποία βρισκόμασταν και τέλος όπως ε, ελέγχθη τα άτομα έχουν μεγάλες δυσκολίες ε, με τις ε, αναφορές τους και αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη η οποία θα προβληθεί διαφορετικά από ό,τι άλλων ατόμων και νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην τηλεόραση πέρυσι που μας έδειχνε τι ε, γίνεται εις ε, το επίπεδο υδατίνων οδών και ε, τι γίνεται με τις κατασκευές στο χώρο αυτό, δωροδοκίες. Η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη και δυστυχώς θα χρειαστεί να παρέμβει η ευρωπαϊκή νομοθεσία διότι βλέπω ότι ε, οι ε, ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν ε, να ξεφύγουν και κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του ότι υπάρχουν άτομα τα οποία παίρνουν παχυλούς μισθούς για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δεν το πράττουν. Κύριε σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς και τη Γραμματεία και τους ε, υπαλλήλου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατανοώ ότι υπάρχει κατανόηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναγνωρίζουμε ε, ότι τους περιορίζει ιδιαίτερα η οδηγία και αν δεν υπάρχει οδηγία δεν υπάρχει εξουσία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Κέλλη, η κυρία Χάρκη και εγώ είχαμε φέρει τρεις οικογένειες που είχαν ε, ε, πρόβλημα και λόγω πιέσεων από εμάς ε, καταφέραμε να λάβουν υποζημιώσεις από τις Ιρλανδικές αρχές. Εξακολουθώ λοιπόν να διατηρώ την ελπίδα ότι κάτι θα προκύψει καλό από αυτή την υπόθεση. Οι πλημμύρες που έπληξαν αυτούς τους ανθρώπους είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που αναφέρουν η κυρία Χάρκιν και ο κύριος Κέλλη ε, ως ο Κέλτικος Τίγρης. Υπάρχουν 95.000 κατοικίες στην Ιρλανδία που δυστυχώς θα πρέπει να ε, να κατεδαφιστούν διότι διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν γίνει σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές. Κατανοώ ότι δεν είναι υπόθεση του Κομισιόν, ε, του Συμβουλίου και ημών, αλλά η Γραμματεία της Επιτροπής Αναφερών θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση βάσει και των επιχειρημάτων που κάναμε η κυρία Χάρκιν και εγώ και κατόπιν να κάνουμε μία πρόταση. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο του 2009 και το τελικό αποτέλεσμα είναι το επιτέλεσμα που επιτύχαμε και μια πολύ ικανοποιητική απάντηση για τις ε, τρεις οικογένειες που έχασαν τις κόρες τους ε, και ε, πριν από κάποια χρόνια, πριν από το 2009 και είναι πολύ ικανοποιημένη. Και ίσως θα έπρεπε η Επιτροπή Αναφοράς να ακούσει τα επιχειρήματά μας και να δει αν υπάρχει περιθώριο ε, ελιγμών. Ε, η οδηγία για τις πλημμύρες δυστυχώς καθυστερεί ακόμα, αλλά πέραν της οδηγίας, αν υπάρχει έστω και ένα ανθρώπινο επιχείρημα που θα μπορούσαμε να προτάξουμε για να μας ακούσουν οι τοπικές αρχές, οι οποίες προφανώς δυστυχώς παραβιάζουν το καθήκον τους και βρίσκονται σε περίπτωση παράβασης καθήκοντος, θα έπρεπε να κάνουν κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποστινάρου. Λίγες παρατηρήσεις. Καταρχάς, όπως μόλις μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του εκπροσώπου της, εδώ δεν υπάρχει σαφής παραβίαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή ευρωπαϊκού κανόνα και αυτό είναι προφανές. Όμως, ένα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, οι δύο κατοικίες κατασκευάστηκαν με οικοδομική άδεια από τις τοπικές αρχές. Επομένως, εδώ υπάρχει νόμιμη κατοικία η οποία σέβεται όλους τους Ιρλανδικούς κανόνες. Δεύτερον, πρόκειται για σαφή ευθύνη των Ιρλανδικών αρχών. Και οι Ιρλανδικέ αρχές είναι οι αρμόδιες για τις άδειε και έχουν δώσει την άδεια για την κατασκευή των δύο κατοικιών. Αυτός που δίνει την έγκριση όμως είναι αυτός ο οποίος ε, έχει και ευθύνε και υποχρεώσεις σε περίπτωση καταστροφής διότι υπήρχαν επιστημονικές εκδείξεις τις οποίες μας αναφέρετε εσείς πριν, υπήρχε ο χάρτης με τις συγκεκριμένες περιοχές ε, επικινδυνότητας πλημμύρας και πού μπορούσαν να κατασκευαστούν κατοικίες και παρόλα αυτά εκχώρησαν άδειες. Εάν λοιπόν υπάρχει τόσο μεγάλο σφάλμα, σαφώς υπάρχει ευθύνη και δεν είναι μόνο πολιτική αλλά ηθική ευθύνη, αλλά υπάρχει νομική ευθύνη. Υπάρχει και η ευθύνη η οποία βαραίνει τους ώμους των τοπικών αρχών που έδωσαν αυτές τις δύο εγκρίσεις. Διότι αν οι δύο πολίτες είχαν κατασκευάσει τις κατοικίες τους χωρίς άδεια, ήταν αυθαίρετες, τότε προφανώς απευθείας θα τους υποχρέωναν να καταβάλουν πρόστιμα. Οι άνθρωποι αυτοί σεβάστηκαν τους κανόνες και τις νομικές απαιτήσεις. Προτείνω λοιπόν ε, στον κύριο Πρόεδρο και τους συναδέλφους καταρχάς να αποστείλουμε μία επιστολή στην Ιρλανδική κυβέρνηση για να ελέγξουμε γιατί δεν ξέρω ακριβώς ε, ε, να πω εδώ ότι δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ιεραρχία σε κάποιες ε, χώρες υπάρχει ειδική υπηρεσία που ασχολείται με τι οικοδομικέ άδειε. Θα πρέπει να ελέγξουμε πώς λειτουργεί το Ιρλανδικό σύστημα και να δούμε αν υπάρχει ευθύνη σε εθνικό επίπεδο και να ελέγξουμε επίσης και ποιο είναι υπεύθυνο σε τοπικό επίπεδο και κατόπιν να αποδοθούν ευθύνε και να ζητήσουμε νομική αποζημίωση για τι δύο αυτέ περιπτώσει. Και μια τελευταία παρατήρηση σε πολλά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται και στη Ρουμανία, όταν ε, ε, πλήττονται από πλημμύρες και, από, και υπάρχουν και καταστρεπτικές συνέπειες από τις πλημμύρες, η κυβέρνηση παρά το γεγονός ότι είναι φτωχός και πολύ αμφίσιμος ο νομικός χώρος που τους επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα, δίνουν κάποιες αποζημιώσεις. Αυτό είναι μια απλή ένδειξη αλληλεγγύης προς ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και εδώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει μόνο ηθική υποχρέωση για τις Ιρλανδικές αρχές, θα πρέπει να συνδράμουν και να δείξουν τη δέωση αλληλεγγύη για τις δύο περιπτώσεις. Διότι οι άνθρωποι αυτοί σεβάστηκαν πλήρως τις νομικές απαιτήσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκονται έρμεα ε, σαν να είχαν κατασκευάσει ε, αυθαίρετες κατοικίες σε ένα κενό χώρο χωρίς καμία νομική διάταξη και χωρίς κανένα σεβασμό των νομικών διατάξεων. Ευχαριστώ πολύ. Please take η κυρία Χάρκιν, θα είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι τα είπαν όλα οι προλαλήσαντες και σας ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, κατανόηση που δείχνουν παρά το γεγονός ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς τους το θέμα και για το γεγονός ότι ε, δέχονται το θέμα και να ευχαριστήσω και τον, ε, κύριο Μποστινάρου για τις καλές του προτάσεις σε κάποιο βαθμό μας περιορίζονται ε, τα όσα μπορούμε να πούμε, αλλά νομίζω ότι μας δώσετε καλές ε, άγουσες. Ε, θα μπορέσουμε ίσως να πιέσουμε λίγο και τις εθνικές κυβερνήσεις για να διασφαλίσουμε πρώτον ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο και δεύτερον να δείξουμε και λίγη κατανόηση για τους ανθρώπους οι οποίοι πλήγησαν από την κατάσταση. Να πω επίσης σε συντομία κάτι για τις ε, τρεις οικογένειες που ήρθαν εδώ για τα οδικά ατυχήματα. Ε, οι οικογένειες αυτές έλαβαν αποζημίωση, αλλά επίσης ε, οι τοπικές αρχές έχουν ενημερωθεί ότι ε, δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη και νομίζω αυτό είναι εισάξιο των αποζημιώσεων να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών και τη Γραμματεία και όλου όσου εξακολουθούν να παρακολουθούν το ζήτημα. Διότι αν δεν το είχαμε συζητήσει εμεί εδώ και το είχαμε αφήσει στη μοίρα του, δεν θα είχαν συμβεί όλα αυτά. Αλλά εσεί το παρακολουθήσατε και βλέπουμε ότι ορισμένε φορέ έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση. Καταρχήν, νομίζω ότι θα αφήσουμε ανοιχτή αυτή την ε, ε αναφορά και ακόμη και αν χρειαστεί να γράψω πολλές επιστολές είναι σαφής η νομική κατάσταση κανονικά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να επέμβουμε πολύ. Ε, έχει, έχει δοθεί η οικοδομική άδεια, έχουν κατασκευαστεί τα κτίσματα και κανονικά η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο επί τόπου. Συμφωνώ ότι στο τέλος οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται αν πρόκειται για δικαστική απόφαση ή για συμφωνία κυρίων. Άρα ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και γι' αυτό θα έλεγα να γράψουμε μία ε, επιστολή, να πούμε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται και να ζητήσουμε να έχουμε μία απάντηση από τις αρχές. Ε, μπορούμε ε, να μπορούμε καταρχήν να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα λάθη τα οποία έχουν γίνει και ε, δυστυχώς ε, δεν ξέρω εάν ε, υπάρχει ένας συνήγορος του πολίτη στην, Ιρλανδία γιατί συνήθως αυτός μπορεί να επέμβει. Άρα ας αφήσουμε ανοιχτό Δεύτερον, να στείλουμε μία επιστολή στις ε, αρμόδιες αρχές εις ε, το, την κυβέρνηση και αν υπάρχει στον συνήγορο του πολίτη. Και στη συνέχεια θα τους πούμε ότι εκφράζουμε την ε, έλλειψη κατανοήσεώς μας διότι ε, αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματα τα οποία έχουν, έπρεπε να έχουν γίνει ε, δεν προχώρησαν. Ωραία. Οπότε αφού συμφωνούμε όλοι κλείνει το σημείο αυτό αλλά έχουμε διάφορα. Έχουμε κι άλλα. Έχουμε το, τα διάφορα τώρα. Λοιπόν, το, ε, τα διάφορα, όπου στα διάφορα έχουμε τα πρακτικά των, ε, της προηγουμένης συνεδριάσεως και στα ε, έχω δύο σημεία, το 20, όπου πρόκειται για την, ε, ε, ε, για την αναφορά 774 της κυρίας Μαρίας Γέζους Χάν από την Ισπανία και όπου θέλαμε να το συζητήσουμε μεταξύ συντονιστών και κατά τη γνώμη μου ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται. Δηλαδή, ε, αγγλικά το ότι ε, θα συζητηθεί στην συνεδρίαση των συντονιστών, δηλαδή θέλαμε να συζητήσουμε και την και το σχέδιο ψηφίσματος θα ήθελα λοιπόν στα πρακτικά να προσθέσουμε αυτό περί ε, σχεδίου ψηφίσματος. Δεν βλέπω κανείς να έχει ε, αντίρρηση και έτσι μπορεί να λήξει η συνεδρίαση αλλά να περιμένουν οι συντονιστές διότι σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση συντονιστών. εγώ θέλω όμως ένα διάλειμμα για 2-3 λεπτά. Θα ψάξω την κυρία Ματσόνη. Εσείς θα μείνετε εδώ μέσα στην αίθουσα. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, δηλαδή στις 5.30.